Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλό σας απόγευμα και ας αρχίσουμε με το πρώτο μας θέμα, δηλαδή την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Το θέμα υπαριθμών 27 για την ανταλλαγή απόψεων, για την προώθηση της ελευθερίας διακίνησης πολιτών και επιχειρήσεων, δια της απλουστεύσεως της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα έχει αναβληθεί. Και το 23 αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου αναβάλλεται επίσης διότι ο ίδιος είναι ασθενής έχετε προτάσεις, ενστάσεις. Κύριε Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Καβαντά. Δύο διευκρινήσεις όσον αφορά τους Ουσπατσίκα. Το πρώτο, η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή μελετούν το ζήτημα, ε, πράγμα που σημαίνει ότι κατά την άποψή μου πρέπει να περιμένουμε τα συμπεράσματά τους. Και το δεύτερο, είναι ότι θα υπάρξουν και κάποιες διευκρινήσεις από τον ίδιο τον κύριο Ούσπατσιτς. Το απόγευμα θα σας, στείλει τις, ε, ε, θα στείλουν τις ε, διευκρινήσεις αυτές που είναι νομικής φύσεως. Επομένως, σας μεταφέρω όλα αυτά τα θέματα όσον αφορά το ζήτημα για την άρση Η κυρία επιθυμώ να τηρήσω τους κανόνες όπως γίνεται και σε άλλες ε, υποθέσεις και αύριο λοιπόν να γίνει η ψηφοφορία για το θέμα του κυρίου Ουσπασκίτς. Τώρα να ζητηθεί ακόμα μία νομική γνωμοδότηση μου φαίνεται ότι δεν είναι αναγκαίο. Έχουμε εξετάσει διεξοδικότατα την υπόθεση αυτή και νομίζω ότι έχει έρθει πια η ώρα η Επιτροπή να λάβει μια απόφαση με ψηφοφορία αύριο. Uh, ο πρόεδρος. Αν κατανοώ καλά είναι διαφορετική η τοποθέτηση των δυο σας για τις δύο διαφορετικές υποθέσεις του κ. Σπάρκητς. Να περιμένουμε, λέει ο κ. Καβατά, να μην περιμένουμε, λέτε εσείς. Άκουσα την άποψη της εισηγητρίας κ. Ρέγνερ. Πράγματι, μου λένε ότι οι νομικέ υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμούν να θέσουν υπόψη μας κάποιες αναλύσεις. Θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να τι θέσω υπόψη σας και μου. Δεν θέλω να επηρεάσω ε, ούτε, τα, ούτε την πορεία διαδικασία, ούτε τα δικαιώματα του ε, προσώπου. Ο πρόεδρος. Να το αφήσουμε λοιπόν για αύριο το πρωί και να δούμε τι θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να το αφήσουμε για αύριο το πρωί. Τι σημαίνει συζήτηση σήμερα ή να το αφήσουμε όπως είχε προβλεφθεί αρχικά. Να το αφήσουμε ως έχει, λέει ο ε, ε, ε, δεν έχω κατανοήσει ακόμη από τη μετάφραση που μου κάνουν λέει ο κ. Καβαντά, όπως προβλέπετε. Ο πρόεδρος, μπορούμε να παρακαλέσουμε τη νομική υπηρεσία αύριο, να τη, να ρωτήσουμε μάλλον αν έχει να παρουσιάσει κάτι. Και σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη να παραμείνει όπως είναι. Αν εσείς κύριε Ρέγνερ. επιθυμώ απλώς να επιβεβαιώσω τα όσα λέτε, ώστε να έχουμε όλοι και τις ίδιες πληροφορίες και να γνωρίζουμε περί τίνο όσα Μιλούμε σήμερα για την ημερήσια, ε, τώρα μάλλον για την ημερήσια διάταξη και αν κατανόησα καλά από αυτά που είπατε κύριε Πρόεδρε, επιθυμείτε να την αφήσετε όπως είναι. Αύριο δηλαδή προβλέπετε αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως και σε αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως θα έχει την ευκαιρία η νομική υπηρεσία να ε, τοποθετηθεί. Ε, είμαι υπέρ αυτής της ιδέας. Πολύ καλά λέει ο κ. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Δύο ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Να σας υπενθυμίσω ότι η κοινή ακρόαση για υψηλό βαθμό λογοδοσίας, διαφάνειας και ακεραιότητας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα διεξαχθεί στις 26 Τρίτου από τις 9 μέχρι τις 12 και 30 στο κτίριο Ζόζεφ Άνταλ στην αίθουσα 4Q2. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις για την ώρα. Το υπαριθμόν 3 που αναφέρεται στην έγκριση των πρακτικών της ε, προηγούμενης συνεδρίασης. Αν δεν λάβω ενστάσεις μέχρι τέλους της συνεδρίασης, τότε θα θεωρήσω ότι τα πρακτικά της 23ης-24ης Δευτέρου θα τα θεωρήσω εγκεκριμένα. Κύριε Πρόεδρε, για την προηγούμενη πρόταση, 26 δεν έχουμε ολομέλη στις Βρυξέλλες. Δεν συμπίπτει η ακρόαση με την ολομέλεια στις Βρυξέλλες, η ακρόαση και τη διαφάνεια που είπατε. Ε, η Ολομέλεια είναι στις 25 Μαρτίου, όχι 26. Περνάμε στο σημείο 5. Την ε, τροποποίηση του καθεστώτος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λόγο έχει ο συγγετής μας ο κύριος Μαρίνιο Πίντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Όταν ανέλαβα την έκθεση, προσπάθησα να εξακριβώσω περί τίνος επρόκειτο διαπίστωσα ότι το πρόβλημα έγκυται στις, ε, στον αριθμό των υποθέσεων. οι αποφάσεις ε, κάθε χρόνο ήταν λιγότερες ε, από τις υποθέσεις που υποβάλλονταν. Έμεναν πολλές υποθέσεις που έμεναν ανεκδίκαστες και μάλιστα δημιουργούνταν μια συσσόρευση χρόνο με το χρόνο εξαιτία τη έλλειψη δικαστών. Υπήρχε ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί. Η πρόταση στην οποία συμπίπταμε όλοι και που υπήρχε από το 2011 ήταν να αυξηθεί ο αριθμό των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου από 28 ε, να αυξηθεί κατά 12. Εγκρίθηκε αυτή η πρόταση αλλά δεν εφαρμόστηκε γιατί το Συμβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει για τα κριτήρια επιλογής και το διορισμό των 12 επιπλέον δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου. Και μάλιστα το Συμβούλιο έπεσε σε αδιέξοδο επειδή το Συμβούλιο παρτίζεται από 28 μέλη, ενώ ο αριθμός των δικαστών που έπρεπε να διοριστούν επιπλέον ήταν 12. Το διέξοδο αυτό κράτησε μία τετραετία, από το 2011. Και η πρόταση που υπευλήθη είναι η αύξηση του αριθμού των δικαστών να μην γίνει μόνο με 12 επιπλέον δικαστές, αλλά με 28, έναν ανακράτος μέλος. Και από τη στιγμή που κάθε χώρα θα μπορούσε να διορίσει έναν επιπλέον δικαστή της ε, δικής της αγένειας, το πρόβλημα θα έβρισκε λύση. Με προβλημάτισε όμως αυτή η πρόταση, γιατί αν αυξάνουμε τον αριθμό των δικαστών από 12 σε 28, δηλαδή διπλασιάσαμε ουσιαστικά το αριθμό των δικαστών. Αυτό δεν το κάναμε ακριβώς για να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά γιατί μόνο με τη, με τη λύση αυτή θα συμφωνούσαν όλα τα κράτη-μέλη και θα προέβαιναν στους ε, διορισμούς. Η τελευταία πρόταση είναι ριζικά διαφορετική. Δηλαδή, αντί για την αύξηση κατά 12 δικαστές, προτείνεται αύξηση κατά 28 και επιπλέον προτείνεται η κατάργηση του Ειδικού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης που προβλεπόταν στις συνθήκες της Νίκαιας και της Λισαβόνας. Οπότε δεν έχουμε μόνο προσθήκη επιπλέον 16 δικαστών, δηλαδή συνολικά διπλασιασμό των δικαστών, αλλά και πρόταση για κατάργηση μιας δικαιοδοσίας ενός δικαστηρίου. Πρόκειται για νέα νομοθετική πρόταση λοιπόν, και μάλιστα μία νέα νομοθετική πρόταση που έχει παρισφρήσει σε μία διαδικασία που είχε ήδη αρχίσει επ' ευκαιρία άλλης νομοθετικής πρότασης. Θεωρώ ότι είναι ασφαλμένη αυτή η διαδικασία. Και με βάση την πορτογαλική ενόμη τάξη, αλλά και θεωρώ ότι με βάση την ενόμη τάξη οποιασδήποτε σύγχρονης χώρας, ε, έχουμε ένα θεσμό που ονομάζεται απάτης βάρος του νόμου. Δηλαδή που προσπαθεί ε, να χρησιμοποιήσει διαδικασίες για να, ε, για να παρακάμψει τον νόμο, για να παρακάμψει κάτι που ο νόμος απαγορεύει ή δεν επιτρέπει. Εμείς με την πρόταση αυτή προσπαθούμε να μεταμορφώσουμε μία νομοθετική πρόταση που στόχο έχει την αύξηση του αριθμού των δικαστών κατά 12, μάλιστα για πρόταση για την οποία έγιναν εκτεταμένες διαβουλεύσεις. Προτείνεται λοιπόν η αύξηση να γίνει όχι μόνο κατά 12 αλλά κατά 28 και επιπλέον προς, προστίθεται η πρόταση να καταργηθεί αυτό το ειδικό δικαστήριο της δημόσιας διοίκησης. Εγώ έχω πρόβλημα με τη νέα πρόταση, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα νομοθετική πρόταση, με νέα πραγματικά περιστατικά. Ζητείτε η κατάργηση ενός ολόκληρου δικαστηρίου. Και οι διαβουλεύσεις που έγιναν ε, το 2011 και το 2012 αφορούσαν μόνο την ανάγκη ή όχι της αύξησης του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου κατά 12. Τώρα όχι μόνο έχουμε περαιτέρω αύξηση, έχουμε από 12 σε 28 και ταυτόχρονα ζητάει και η κατάργηση του δικαστηρίου της δημόσιας διοίκησης. Κανένας όμως δεν έδωσε τη γνώμη του ούτε για την επιπλέον αύξηση του αριθμού των ε, δικαστών, ούτε για την πρόταση κατάργησης του ειδικού δικαστηρίου. Αυτή είναι βέβαια και η μοναδική λύση που έχει υποβληθεί μέχρι τώρα. Και, είναι και η πιο δαπανηρή, η πιο επαχθής λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα για τους ε, φορολογούμενους. Γιατί κάθε δικαστή ε, κοστίζει το χρόνο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε τέτοιου είδου επαχθεί ε, προτάσει, ε, τόσο δαπανηρέ, πώ θα την προβάλλουμε και πώ θα την υποστηρίξουμε στην κοινή γνώμη, ενώ ζητούμε από πολλέ χώρε δραστικέ περικοπέ των δημοσίων δαπανών και σε χώρε όπω η δική μου επιβλήθηκαν δρακόντια μέτρα λιτότητας. Και τώρα εμεί δεν συμφωνούμε να διοριστούν μόνο 10 επιπλέον δικαστέ, να διοριστούν επιπλέον 28. Νομίζω δεν μπορούμε. Από τη μια να ζητούμε τόσε θυσίε από του ε, Ευρωπαίου φορολογούμενου και εμεί αυξάνουμε έτσι τον αριθμό των δικαστών. Επίση, ε, δεν έγινε σωστή ανάλυση των προβλημάτων. Γιατί, γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμό των υποθέσεων του κάθε δικαστή. Γιατί δεν απλουστεύεται η δικονομική διαδικασία ώστε να εκδικάζεται πιο γρήγορα μια υπόθεση. Γιατί δεν προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να κάνει μια προκαταρκτική αξιολόγηση του παραδεκτού ή όχι των ε, συγκεκριμένων υποθέσεων. Γιατί στις Ηνωμένε Πολιτείες το ανώτατο δικαστήριο κρίνει μη παραδεκτές ορισμένες υποθέσεις. Το ίδιο γίνεται και στην Πορτογαλία μπορεί προδικαστικά να κληθούν παραδεκτέ ε, κάποιε υποθέσει. Ακόμη και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει τέτοιε διαδικασίε. Γιατί τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να μην έχουν τέτοιε προκαταρκτικέ διαδικασίε και να γίνεται μια νομικοτεχνική αξιολόγηση του εφικτού τη υπόθεση και του παραδεκτού, για να μην φτάνει στα δικαστήρια και να μειώνεται το άχθο των δικαστών. Επίση, ε, γιατί να μην έχουμε ένα βραβείο παραγωγικότητα των δικαστών, γιατί η παραγωγικότητα του δικαστή αφορά τον αριθμό των υποθέσεων που εκδικάζει σε μία δεδομένη περίοδο. Σήμερα μιλάμε παντού για παραγωγικότητα. Ποια είναι όμως η, το αντικειμενικό κριτήριο της παραγωγικότητας για έναν δικαστή του ΔΕΚ, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινότητων, γιατί ένα δικαστή πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στην Πορτογαλία εκδικάζει πάνω από 400 υποθέσει το χρόνο. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάθε χρόνο εκδικάζονται περίπου 90.000 υποθέσει υποθέσεις για 47 δικαστέ. Στην Πορτογαλία το Πορτογαλικό Συνταγματικό Δικαστήριο εκδίκασε 1.700 υποθέσεις μόνο το 2014. Και οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κάθε ένας από αυτούς εκδικάζει λιγότερο από 25 υποθέσει το χρόνο. Εντάξει, μπορεί να είναι πιο περίπλοκες ε, υποθέσεις, αλλά δεν ισχύει πάντα αυτό. Γιατί είναι τόσο χαμηλός ο αριθμός των ε, ε, εκδικαστησών αποφάσεων από τους Ευρωπαίους δικαστές. Μπορούμε να θεσπίσουμε κάποια αντικειμενικά κριτήρια παραγωγικότητας, γιατί η παραγωγικότητα είναι βασικό κριτήριο για κάθε εργαζόμενο. Από το, από το κάθε εργοστάσιο μέχρι το κάθε ε, κοινοτικό θεσμικό όργανο πρέπει να κρίνεται η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα κάθε εργαζομένου. Αυτό ισχύει για όλους μας για τον κάθε εργάτη, για τον κάθε μισθωτό, για τον κάθε δικαστή. Γιατί να μην έχουμε τέτοια κριτήρια παραγωγικότητας. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε το ίδιο απαιτητικοί από τους αυτούς μας όσο είμαστε και από τους υπόλοιπους. Γιατί λοιπόν να μην θεσπίσουμε τέτοια κριτήρια παραγωγικότητας και για τους δικαστές. Βέβαια κάτι τέτοιο προϋποθέτει μελέτες επιπτώσεων. Πρέπει να γίνουν σωστές τεκμηριωμένες μελέτες, άρτιες, για να δούμε πού οφείλεται αυτή η κατάσταση και αυτή η συσσόρευση υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης, στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα καμία ακρόαση με οποιοδήποτε δικαστή του Γενικού Δικαστήριου. Δεν είχαμε ευκαιρία να μιλήσουμε ούτε με ένα δικαστή του Γενικού Δικαστήριου. Γιατί, γιατί, γιατί το πρόβλημα το έχουμε με το Γενικό Δικαστήριο. Το Γενικό Δικαστήριο παρουσιάζει τέτοια ολιγορία στην εκδίκαση των υποθέσεων και έχουμε τέτοια συσσόρευση υποθέσεων. Γιατί δεν ακούσαμε ούτε μία φορά ένα δικαστή να έρθει εδώ και να μα εξηγήσει πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση που υποβάλλω. Να οργανώσουμε συνομιλίε και ακροάσει με δικαστέ του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Να καλέσουμε και τον πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου για να μα πει τι συμβαίνει, πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση. Νομίζω ότι έτσι θα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Να δούμε πού έγκυται το πρόβλημα και να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών, να αυξήσουμε τον αριθμό των προδικαστικών ζητημάτων, να προβλέψουμε ένα βραβείο επιδόσεων παραγωγικότητας. Να καθορίσουμε και ένα νομικό έπαθλο για τους πιο παραγωγικούς ε, δικαστές. Αυτούς που ξεπερνούν δηλαδή το μέσο όρο των ε, εκδικαστικών υποθέσεων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ε, κρίνουμε με βάση πληροφορίες που λαμβάνουμε από δεύτερο και τρίτο χέρι. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε ένα βήμα και να ακούσουμε από πρώτο χέρι, από τον άμεσα ενδιαφερόμενο το πρόβλημα, από τους ίδιους τους δικαστές δηλαδή του Γενικού Δικαστηρίου. Μάλιστα έλαβα γνώση ενός ε, εγγράφου που το έχουν προσυπογράψει όλοι οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου και κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2014. Και μάλιστα οι, οι δικαστές είναι κατά της πρότασης που συζητούμε. Βλέπετε ότι στο έγγραφο που προσπέγραψαν όλοι οι δικαστές είναι κατά της πρότασης. Γιατί δεν έφτασε αυτό το έγγραφο με την αρνητική γνώμη των ίδιων των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο πρόεδρος του, Ευρωπαϊκού, του Γενικού Δικαστηρίου και όλοι οι δικαστές υπέγραψαν αυτό το έγγραφο στο οποίο αποφαίνονται κατά της πρότασης. Γιατί δεν έφτασε επίσημα αυτό το έγγραφο στην Νομική Επιτροπή, γιατί δεν έφτασε επίσημα αυτό το έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμένα μου το έστειλαν προσωπικά. Έτσι το κοίταξα και είδα τι έλεγε. Γιατί αν ισχύει όντω αυτή η αντίθετη γνώμη του δικαστηρίου, τι κάνουμε εδώ. Τι παίζουμε τον Καραγκιόζη, θέατρο σκιών. Το ίδιο το Γενικό Δικαστήριο λέει το πρόβλημα δεν θα λυθεί με την αύξηση των δικαστών, αλλά με την καλύτερη, ε, με την αύξηση του αριθμού των προδικαστικών ε, διαδικασιών. Γιατί λοιπόν δεν έφτασε αυτό το έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συγκεκριμένη αρμόδια επιτροπή, την νομική επιτροπή. Αυτό διερωτώ γιατί είναι πολύ σημαντικό έγγραφο. Επίσης, έμαθα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου απειλήθηκε. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε εις βάρος του πειθαρχική διαδικασία ή απλώς άκουσε, υπήρχε απειλή τέτοιας έναρξης ε, πειθαρχικής διαδικασίας ακριβώς επειδή υπέγραψε μαζί με τους συναδέλφους του το σχετικό έγγραφο. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να λάβουμε επίσημη απόφαση σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Εγώ θα ήθελα και πιστεύω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκπαιρεώσω το έργο μου και να εκπονήσω την έκθεση, να ακούσουμε τη γνώμη των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου για να δούμε τι έχουν να μας πούν. Γιατί μιλούμε για δικαστές. Οι δικαστές έχουν την ίδια αξιοπρέπεια, είτε ε, είναι δικαστές πρωτοβάθμιου δικαστηρίου είτε δικαστές ανωτάτου δικαστηρίου, αρίου πάγου ή συνταγματικού δικαστηρίου. Και το πρωταρχικό σημείο σε κάθε σύγχρονο κράτος δικαίου είναι η ανεξαρτησία του δικαστή. Θα πρέπει να βρίσκεται στο απειρόβλητο οποιασδήποτε επιρροής ο δικαστής. Και μάλιστα η ανεξαρτησία του θα πρέπει να είναι όχι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική ε, θα πρέπει ο κάθε δικαστή και στο όργανο που υπηρετεί τη θητεία του να είναι ανεξάρτητο και να μην υφίσταται καμία πίεση, καμία απειλή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο έργο του. Αυτά λοιπόν. Έχουμε έγγραφο που έχει υπογράψει ο πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου και όλοι οι δικαστές του και που ε, λαμβάνουν θέση κατά τις θέσεις, ε, τις πρώτες που έγινε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερες μελέτες και κυρίως μια μελέτη επιπτώσεων των επιμέρους προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λυθεί το πρόβλημα. Οπότε, η συγκεκριμένη μου πρόταση είναι να καλέσουμε τους δικαστές. Θα ήθελα εσείς κύριε Πρόεδρε να υποβάλλετε ένα κατεπήγον αίτημα για διεξαγωγή ακρόασης, δημόσιας ακρόασης με τον πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου και με δικαστές για να δούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να εμποδίζουμε τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών να μάθουν από τα χίλια του ίδιου του ενδιαφερομένου που έγκυται το πρόβλημα και τι γίνεται με το Γενικό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χαουτάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πρέπει να πω ότι με προβληματίζει ε, που βλέπουμε οικονομικά αυτό το ζήτημα. Στην ε, ίδια μου τη χώρα είδα ότι οι περικοπές και τα ε, μέτρα τα οικονομικά τα οποία ελήφθησαν είχαν πολύ κακό αποτέλεσμα επί του νομικού συστήματος και ενδεχομένως μπορούν να προκύψουν καταστάσεις όπου όντως ε, η, ε, ε, η επιβραδυμένη πρόσβαση να είναι στην ουσία άρνηση απόδοσης σε δικαιοσύνης. Εν πάση περιπτώσει λέμε ότι ο κάθε ένας ευρωβουλευτής κοστίζει 60% από ότι ο δικαστής ε, και επομένως τι λέτε, λέτε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε ας πούμε να μειώνουμε τον αριθμό των ευρωβουλευτών έτσι ώστε να, ε, μέσω περικοπών να κερδίσουμε οικονομικά και από εκεί. Ίσως τότε προκύψει μια κατάσταση όπου ε, πραγματικά θα είναι υπορφορτωμένο το δικαστήριο, η παραγωγικότητά τους δεν θα είναι καλή Κατά την άποψή μου νομίζω και από όσα γνωρίζω ε, νομίζω ότι το Γενικό Δικαστήριο πέρυσι αποφάσισε ε, επί 800 ε, υποθέσεων και έμειναν απ' έξω 900 και από όσο ξέρω 2 με 3 χρόνια διαρκεί η διαδικασία για κάθε υπόθεση και αυτό είναι πραγματικά υπερβολικά πολύ. Είχα την δυνατότητα να συζητήσω με δικαστές, όπως και άλλοι συνάδελφοι, όταν ε, κόπηκε το μικρόφωνο της ομιλητρίας, όταν ε, ε, πήγαμε στο δικαστήριο. Έχω την εντύπωση ότι ήδη το δικαστήριο αλλάζει τις εσωτερικές διαδικασίες και ενδεχομένως προβλέπει και κάποια δικαστικά τέλη για, τις, για όσους μπορούν να τα πληρώσουν. Επομένως είναι γεγονός ότι και οι ίδιοι παίρνουν το θέμα πολύ στα σοβαρά σε ορισμένα χρόνια ενδεχομένως φοβούμε ότι ε, θα ε, υπάρχει τόσο βεβαρημένο πλέον πινάκιο που ε, δεν θα ξέρουμε πώς να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ήδη, ήδη τώρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο Μηνίων έχει ζητήσει κάποια αντισταθμίσματα ακριβώς λόγω της βραδύτητας με την οποία αποδίδεται η δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τώρα, εάν, εάν δεχτούμε την απόφαση ε, διπλασιασμού του αριθμού των δικαστών, ε, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο ε, και προηγούμενες αποφάσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ισότητα των φύλων και νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι εάν θα έχει κάθε χώρα δύο δικαστές θα πρέπει να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτή την πρακτική της ισότητας των φύλων και σας ξαναλέω λέω συνάδελφοι ότι ήδη έχουμε πάρει ε, τέτοιου είδου θέσει. άρα μόνο θα ευθυγραμμιστούμε με τις προηγούμενες αποφάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Σβιεύκα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η προηγούμενη πολύ σημαντική και ε, συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση με πρόεδρο της ε, Λατωνικής Προεδρίας. Υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία. Εντάξει τώρα. Επαναλαμβάνω, η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με την ε, Λετωνική Προεδρία με οδήγησε στο συμπέρασμα να σκεφτώ που κάναμε το λάθος. Κάναμε το λάθος ε, στη μεταρρύθμιση ε, του ΔΕΚ. Γιατί με τη μεταρρύθμιση αυτή ασχολούμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε σε αυτό το θέμα. Είχαμε πολλές συναντήσεις. Είχαμε συναντήσεις ε, με τον πρόεδρο του δικαστήριου, τον κύριο Σκουρή. Είχαμε συναντήσει με του δικαστέ του Γενικού Δικαστηρίου. Και σε κάθε ε, συζήτηση το συμπέρασμα ήταν το ίδιο το δικαστήριο πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπό αυτό το πρίσμα, υπό αυτό το πυλώνα, κρίνουν οι πολίτε και οι επιχειρηματίε κατά πόσο λειτουργεί σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με την περαιτέρω αναβολή τη απόφαση για τη μεταρρύθμιση, γιατί χρονοτρίβησε υπερβολικά το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν έτοιμο από κοινού με το δικαστήριο, γιατί είχαμε σύντοση απόψεων και με τον πρόεδρο Σκουρή και με του δικαστέ για την αναγκαιότητα τη μεταρρύθμιση. Και ε, εκπλήσωμε και με την ε, πληροφορία του εισηγητού ότι υπήρχε ένα μυστικό έγγραφο στο οποίο βλέπουν, λένε οι δικαστές ότι διαφωνούν. Το θέμα είναι να δούμε σε τι διαφωνούν και με τι μέθοδο διαφωνούν. Γιατί ε, προτείνονται και άλλες μέθοδοι και άλλες προτάσεις. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος Κουρίς είχε πει ε, κατηγορηματικά ότι κάθε μεταρρύθμιση του δικαστηρίου που ε, θα βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του θα γίνει δεκτή από το δικαστήριο. Και θέσαμε πέντε ερωτήσεις και λάβαμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε, την, έχουμε λάβει την επιστολή του Προέδρου Σκουρί και σε αυτή την επιστολή φαίνεται καθαρά και εξάστερα ποια είναι η κατάσταση, η σημερινή κατάσταση, η τραγική σημερινή κατάσταση στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Γιατί αναφέρθηκε το οικονομικό ζήτημα και μου άρεσε πολύ αυτό που είπε πριν από λίγο η κυρία Χάουταλα. Ότι αν είναι υπερβολικό το κόστο του δικαστηρίου, είναι υπερβολικό το κόστο του και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α το σκεφτούμε λίγο. Λέμε ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών επειδή κάτι τέτοιο θα είναι δαπανηρό για τον προπολογισμό. Ξέρετε τι πρόστιμα ε, πρέπει να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστερήσεις της εκδικάσεις είναι δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες ε, εκατομμύρια. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η αύξηση του αριθμού των δικαστών. Μιλάμε για το οικονομικό θέμα, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον ζήτημα. Η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης είναι σημαντική. Ε, βέβαια, με βάση την ε, συνθήκη της νίκης προτείνεται διτή λύση είτε μέσω της αύξησης του αριθμού των δικαστών είτε μέσω της ε, δημιουργίας ειδικών δικαστηρίων. Αν υιοθετήσουμε την αύξηση του αριθμού των ε, δικαστών και όχι την, αριθμό των οδικών δικαστηρίων, το αποτέλεσμα είναι σαφές ο μοναδικός, το μοναδικό ειδικό δικαστήριο που είναι το δικαστήριο Δημόσια Διοίκηση είναι, φαίνεται ένα δικαστήριο που δεν είναι αποτελεσματικό, είναι τελείως αναποτελεσματικό γιατί οι δικαστέ που απασχολούνται εκεί δεν έχουν πολλέ υποθέσει να εκδικάσουν. Δεν μπορούμε όμω να του πούμε α, ότι θα πρέπει να, αναφέρ, να, να λάβετε τα θέματα του Γενικού Δικαστηρίου. Μένουν λοιπόν πολλοί δικαστέ αναξιοποιητοί στο ειδικό δικαστήριο δημόσια Διοίκηση. Το καλύτερο λοιπόν είναι να αφήσουμε τον αριθμό των δικαστών, όχι να έχουμε ειδικό δικαστήριο. Επίσης, το θέμα της πρόσληψης ηγητών, όχι οι δικαστές. Ποιος όμως θα εκδικάσει το θέμα, οι γραμματεί, οι συγητές, οι βοηθοί, όχι οι δικαστές. Ο εισηγητής θα αποφασίσει για την εκδίκαση της υπόφασης, της ε, δικαστικής απόφασης. Γιατί το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για θέματα που έχουν ε, δικογραφία και 100.000 σελίδων μερικές φορές. Ποιο θα διαβάσει όλα αυτά, ο γραμματέας, ο εισηγητής. Δεν μπορεί ένα εισηγητή με τέτοια ε, ογκοδέστατη, ένα δικαστή με ένα τέτοια ογκοδέστατη δικογραφία να εκδικάζει σοριδών αποφάσει. Ούτε να τα αναθέσει όλα στον εισηγητή. Θα πρέπει για να εξοικειωθεί με την ουσία τη υπόθεση ένα δικαστή ε, να έχει χρόνο στη διάθεσή του. Γιατί οι υποθέσει είναι πολύ δύσκολε και περίπλοκε πολλέ φορέ. Και για να πετύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του Γενικού Δικαστηρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών. Τώρα, για απόφαση προδικαστική για θα πρέπει να φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο. Πόσε τέτοιε υποθέσει είχαμε, πόσε υποθέσει είχαμε που το δικαστήριο απέρριψε αποφάσει, ε, απέρριψε υποθέσει α μη παραδεκτέ. Ελάχιστε καθόλου. Α μην λοιπόν καταθέτουμε προτάσει που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επίση, η διαδικασία είναι δυναμική. Γι' αυτό και στη διάρκεια τη υποβλήθηκαν πολλέ προτάσει. Ε, στην αρχή είπαμε πώς θα βρούμε τους επιπλέον 12 δικαστές. Εμείς ε, που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήσαμε αρχικά να πούμε όχι τώρα διαφωνούμε με την αύξηση του αριθμού των δικαστών. Δημιουργήθηκε μία απέλπιδα και ανόητη κατάσταση. Ε, και αυτή την εντύπωση θα δώσουμε, ότι στην αρχή να πούμε ναι συμφωνούμε με την αρχή, με την αρχή της αύξησης των δικαστών και τώρα λέμε όχι. Πολύ πρόσφατα πραγματοποίησαμε επίσκεψη στο Λουξεμβούργο. Συναντηθήκαμε με προέδρους όλων των δικαστηρίων, όλων των βαθμών. Είχαμε συναντήσεις με δικαστές και όλες οι συζητήσεις κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Μεταρρύθμιση αμελητή, πάρα αυτά, το συντομότερο δυνατό. Μεταρρύθμιση στην οποία θα συμφωνήσουν όλοι. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και το ίδιο το Δικαστήριο. Και έχουμε επιτέλους μία πρόταση που μας ε, φέρνει πιο κοντά στην αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων. Δεν θα πρέπει το κοινοβούλιο αυτή τη φορά να αποτελέσει τροχοπέδι σε αυτή τη μεταρρύθμιση που είναι απαραίτητη και το γνωρίζουμε κάλλιστα ότι είναι απαραίτητη. Αν κάποιο δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη τη μεταρρύθμιση, α ρωτήσει και θα του απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να προκαταλάβω τα όσα θα πει η σκιώδη συγκεντριά μας, θα τα αναπτύξει μόνη της, αλλά χαίρομαι για τα όσα είπε και ο Σβιεύκα και η κυρία Χαόταλα. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι απόλυτα αναγκαία. Ήδη μας απασχολεί πολύ καιρό και δεν θα πρέπει να αναβληθεί περισσότερο. Γιατί άραγε. Είχε, υπήρξε ευκαιρία για να τοποθετηθούν και οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν είναι ο μέγας άγνωστος η θέση των Ευρωπαίων δικαστών, τα επιχειρήματά τους είναι γνωστά. Να μου επιτρέψετε να έλθω σε δύο θέματα. Αφενός, ας το πω έτσι ε, απλοϊκά, αυτό το επίδομα είναι όμως πάρα πολύ διαφορετικές υποθέσεις. Άλλες, ε, ε, άλλες υποθέσεις είναι τεράστιες, άλλες είναι πολύ πιο μικρές και απλές. Δεν μπορεί να τα εξετάσει και να, να αυτά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Σε μια δημοκρατία είναι απόλυτα απαραίτητο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στην δικαιοδοτική εξουσία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το δικαστήριο, γι' αυτό χρειαζόμαστε και τα στοιχεία που έχουν αναφέρει οι συγητές οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ασφαλώς και είχαν ευκαιρία να τοποθετηθούν, να υποβάλουν τα επιχειρήματά τους. Τα έχουμε συζητήσει αυτά κατά επανάληψη. Και ιδίω τώρα, ενώ του γεγονότος ότι το Συμβούλιο αναπτύσσει μια τελείω διαφορετική δυναμική. Πρέπει λοιπόν η διαπραγμάτευση να καταλήξει κάπου επικοδομητικά και όχι να ξανανοίξει ολόκληρη δέσμη. Κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί. Euh, le Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ε, δικαστήριο και ε, ε, και πρωτοδικείο που να λειτουργούν ε, σωστά ε, και, και να είναι η πρόσβαση προς την δικαιοσύνη σωστή για όλους τους πολίτες, μια δικαιοσύνη η οποία θα λειτουργεί ε, σε σωστά χρονικά όρια. Ένα έγκριτο νομικό θα έπρεπε να ξέρει ότι είναι δύσκολο να μετρήσει κανεί την παραγωγικότητα ενό δικαστηρίου όπω είναι το 10 δεν ε, τολμώ να εκφραστώ όσον αφορά την παραγωγικότητα των βουλευτών ή πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε την παραγωγικότητα αυτή. Απ' την άλλη πλευρά, μετά από πολλές συζητήσεις που είχαμε με τους ε, δικαστές και του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου, Φαίνεται ότι αν θέλουμε να αυξήσουμε την ε, παραγωγικότητα των ε, ε, δικαστών, ίσως καλό θα ήταν να επιμηκυνθεί η θητεία τους, γιατί την πρώτη χρονιά μόλις φτάνουν πρέπει να μάθουν λίγο τον τρόπο λειτουργίας και τα θέματα και το τελευταίο χρόνο της θητείας τους δεν δέχονται πλέον καινούργιες υποθέσεις, γιατί δεν θα έχουν το χρόνο να τις αντιμετωπίσουν. Επομένως, ενδεχομένως θητείες πιο μεγάλες, έτσι ώστε να είναι ε, μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα ή βελτιωμένη η αποτελεσματικότητα. Δύο λόγια όσον αφορά τη μεταρρύθμιση. Κατά την άποψή μου δεν έγινε λόγος ε, για μεταρρύθμιση. Ε, απλώς συζητήσαμε την ανάγκη αύξησης του αριθμού των δικαστών. Το Κοινοβούλιο βρήκε το 2014 μία συμφωνία έτσι ώστε να γίνουν 12 οι δικαστές τότε όλοι συμφωνούσαν ότι θα έπρεπε κατά 12 να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών αλλά χάλασαν τα πράγματα στις συζητήσεις στο Συμβούλιο γιατί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ε, οι χώρες όσον αφορά τον διορισμό των δικαστών. Και αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερο λυπηρό. Εάν οι χώρε μέλη είχαν επιτύχει συμφωνία, δεν θα ξανασυζητούσαμε σήμερα εδώ το θέμα. Δεν ξέρω βέβαια πώ μπορούν να πιστούν να είναι πιο λογικά τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια άλλη πρόκληση που θα έχουμε μπροστά μα. Έχω την εντύπωση μετά από τις συζητήσεις ε, που είχα επισήμως και ανεπισήμως με κάποιους δικαστές, έχω την εντύπωση, λέω, ότι η πρόταση ε, είναι πραγματικά η τελευταία ε, δυνατότητα και γιατί από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να αυξήσουν κατά 12 αποφάσισαν να διπλασιάσουν τον αριθμό των δικαστών ε, και νομίζω ότι αυτό και θα συμφωνήσουν και άλλοι μαζί μου ότι ε, αυτό σαν κίνηση είναι υπερβολικό αλλά βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο για να δούμε αν και κατά πόσον μπορούν να ικανοποιηθούν με τον μικρότερο αριθμό, με τα 12 μέλη. Αλλά βέβαια ο κύριος Ζεύκα προηγουμένως ε, σωστά αναρωτιέται ε, θα πρέπει να τα μπλοκάρουμε όλα γιατί ε, διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την πρόταση, θεωρώντας ότι πραγματικά δεν είναι η εξαιρετική πρόταση, αλλά ε, τι να σας πω, εάν θυμάστε την πρόταση του Προέδρου του Δικαστηρίου προτείνει σε μία πρώτη φάση να, ο αριθμός να φτάσει στους 12, μετά ε, να ε, καταργηθεί το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και να ενσωματωθεί με το ε, Πρωτοδικείο και μετά να συνεχίσουμε. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι ε, ε, δεν φανταζόταν ότι θα σταματήσουμε στην πρώτη φάση, γιατί η πρώτη φάση είναι η εξέβρεση μιας συνένεσης. Ε, άρα θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα τοποθετηθούν τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα που είναι πραγματικό, δηλαδή η λειτουργία του πρωτοδικίου και του 10 και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση και τις αναλύσεις από την αρχή. Έγιναν, ξανά έγιναν στο παρελθόν και Πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει ε, να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών. Εγώ λέω ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ε, προς τη λύση δηλαδή του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας ε, την αγαπητή συνάδελφη Ντελβό, ανερωτιόμουν εάν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μια τεχνική με πάρε ε, Δηλαδή, ε, χρειάζεται για την καλή του λειτουργία το δικαστήριο περισσότερους δικαστές και να πούμε ότι εμείς θα δούμε το θέμα ευνοϊκά εάν εσείς Συμβούλιο, γιατί στο Συμβούλιο συζητιέται το θέμα, εσείς Συμβούλιο μας δώσετε σαν αντάλλαγμα την ε, ε, επιμήκυση της θητείας. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο σύντομες οι θητείες. Αναρωτιέμαι γιατί οι ε, κυβερνήσεις θέλουν να ευχαριστήσουν περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να, βάλουμε, να εφαρμόσουμε ένα σύστημα όπου ο ένας δίνει και ο άλλος επιστρέφει κάτι σε αντάλλαγμα έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια δικαιοσύνη η οποία να λειτουργεί καλά γιατί αυτή ακριβώς η δικαιοσύνη είναι ένας πυλώνας πολύ σημαντικός για τους πολίτες και το να περιμένει ένας πολίτης επίλυση του ζητήματος του δύο και τρία χρόνια δεν είναι λογικό. Ευχαριστώ. Ε, Συμφωνεί η ομάδα μας ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού μηχανισμού της Ένωσης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι είδους μεταρρύθμιση. Η απλή αύξηση του αριθμού των δικαστών δεν απαντά στο πιο σοβαρό πρόβλημά μας. Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε ένα έλλειμμα δικαστικής προστασίας καθώς και σε δεύτερο βαθμό που υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού, ε, της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και τον ίδιο τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη, κάτι που έχει να κάνει πρώτα με τη δυνατότητα να υποβάλλονται ένδικα μέσα, ιδίως στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αλλά και βεβαίω και εγγύησης ανεξαρτησίας των δικαστών που συναπαρτίζουν το δικαστήριο. Για το πρώτο, πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ιδίως για τα συνδικάτα και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε αυτές να μπορούν να αμφισβητήσουν την ισχύ και νομιμότητα διαφόρων μέτρων που θεσπίζει η ίδια η Ένωση, είτε το Συμβούλιο Υπουργών, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το δεύτερο πρόβλημα, πρέπει να ενισχύσουμε τις εγγύησεις δικαστικής ανεξαρτησίας σε επίπεδο τουλάχιστον ισότιμο εκείνου του, των εχεγγύων δηλαδή ανεξαρτησίας των δικαστών του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα, όχι επαναδιορισμοί, να απαγορεύονται απολύτως. Επίσης, η διαδικασία διορισμού να ομοιογενοποιηθεί, να είναι ομοιογενής δηλαδή, σε όλες τις χώρες και να είναι προσαρμοσμένη τουλάχιστον στις απαιτήσει που ισχύουν για τους δικαστές του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπερψηφίσουμε η ποτέ αύξηση του αριθμού των δικαστών είτε του πρώην πρωτοδικειου είτε του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ούτε θα δεχθούμε καμιά αύξηση αριθμού δικαστών μέχρι ότου υπάρξουν μέχρι ότου ενισχυθούν οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας μέσα από αναθεώρηση των συνθηκών. Mrs. Hautala. Κύριε Χάουταλα. Κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω κάποιες πληροφορίες. Οι νέοι οργανισμοί επίσης θα οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των εισερχομένων υποθέσεων. Υπάρχει ανησυχία ότι για παράδειγμα ο οργανισμός για τα χημικά θα αρχίσει να προκαλεί υποθέσεις και επομένως ακόμα μεγαλύτερος φόρτος εργασίας για το δικαστήριο και υπάρχουν και παραπάνω από 100 υποθέσεις που έχουν σχέση με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτό που προσπαθώ να πω λοιπόν με λίγα λόγια είναι ότι ίσως το 2011 όταν ανέκυψε για πρώτη φορά το θέμα με αριθμό για αύξηση των θέσεων των δικαστών 12 αλλά βασισμένο στον τότε αριθμό των υποθέσεων πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και προς τα εμπρός στο μέλλον πώς εξελίσσεται ο φόρτος εργασίας και γι' αυτό αυτός ο αριθμός 28 δεν μου φαίνεται αδικαιολόγητος. Κύριε Μαρίνιο Επίντου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από όλα όσα ακούσαμε, αντλώ το συμπέρασμα ότι δημιουργείται επιτακτική ανάγκη ρηξικέλθης μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δικαιοσύνης. Θέλουμε μια δικαιοσύνη και μια μεταρρυθμίση που θα ενισχύει την ανεξαρτησία των δικαστών, ιδιαίτερα απέναντι στην πολιτική εξουσία. Γιατί ένας δικαστής που μπορεί να διοριστεί από οποιονδήποτε, από αρχή γίνεται, πολύ δύσκολα θα ασκήσει τουλάχιστον την πρώτη θητεία ανεξάρτητα. Γιατί θα προσπαθήσει να επιστρέψει ε, τη χάρη προς την αρχή που τον διόρισε, ε, ευελπιστώντας ότι θα ξαναδιοριστεί. Από εμπειρίες που είχαμε και με άλλα δικαστήρια, το Πορτογαλικό ε, Συνταγματικό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ήταν να ήταν η παράταση της αρχικής θητείας χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, επαναδιορισμού. Ε, φαίνεται ότι οι αντιδράσεις στην αρχική μου ε, παρέμβαση με οδηγούν στο εξή συμπέρασμα. Αν γίνει δεκτή η πρόταση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το Γενικό Δικαστήριο θα βρεθεί με 56 δικαστές ε, κάθε έχει 25 ε, υποθέσεις από τις χίλιες υποθέσεις που λαμβάνει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 47 δικαστές για 90.000 υποθέσεις που εκδικάζει κάθε χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να πω στην συνάδελφο Ντελβό ότι κανείς δεν πρέπει να φοβάται την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα είναι κριτήριο αξιολόγηση το οποίο θα πρέπει όλοι να υπαγόμαστε. Είτε είμαστε πολιτικοί, είτε είμαστε πρόεδροι δημοκρατίας, είτε είμαστε βουλευτές, είτε είμαστε δικαστές. Η παραγωγικότητα είναι το κριτήριο αξιολόγηση οποιοδήποτε εργαζομένου. Εγώ ως βουλευτής δεν φοβάμαι να αξιολογηθώ με βάση το κριτήριο της παραγωγικότητας. Μάλιστα, θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να σας πω ότι εγώ Είμαι αποκλειστικά ευρωβουλευτής, είναι η μοναδική μου αρμοδιότητα και όταν ανέλαβα το κοινοβουλευτικό μου έργο παραιτήθηκα από δικαστής γιατί θεωρώ ότι είναι ε, ασύμβατο σε, μία, σε ένα όργανο να νομοθετεί κανείς και, σε, και αλλού να είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή αυτών των νόμων. Ούτε έχω ε, πελάτες ιδιώτες που ενδιαφέρονται για την νομοθεσία που θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι αποκλειστικά και μόνο Ευρωβουλευτή. Και δεν φοβάμαι καθόλου την παραγωγικότητα. Και όταν μιλώ για απώλεια παραγωγικότητα του δικαστή, είναι γιατί μειώνεται ο αριθμό, ο μέσο ε, αριθμό των ε, δικαστησών υποθέσεων. Οι Πορτογάλοι δικαστέ εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούν ακριβώ ε, την το κριτήριο τη παραγωγικότητας. Θέλω για κάθε δικαστή να αναφέρει το αριθμό των υποθέσεων που εκδικάζει κάθε χρόνο. Γιατί να μην έχουμε τέτοιου δείκτες και για τι υποθέσεις που εκδικάζει το Γενικό Δικαστήριο. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2015 κατατέθηκαν 127 υποθέσεις στο Γενικό Δικαστήριο. Εκδικάστηκαν 200 υποθέσεις μόνο επειδή ο αριθμός των νέων εισηγητών είχε αυξηθεί. Δηλαδή, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2015, το Γενικό Δικαστήριο έλαβε αποφάσεις για 70% το 100 των αποφάσεων. Αυτή είναι η καλή λύση, αυτή είναι, αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Γιατί μας δίνει την εντύπωση ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος και λιγότερος, λιγότερο προσωπικό. Και είπατε ότι το Συμβούλιο αν θέλει να αποφασίσει τον αριθμό των δικαστών. Μα δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου η απόφαση για την αύξηση του αριθμού των δικαστών. Υπάρχει συναπόφαση για το θέμα αυτό. Ισχύει συναπόφαση. Θα συναποφασίσουμε με το Συμβούλιο θα πρέπει και εμείς να συμφωνήσουμε με την αύξηση του αριθμού των δικαστών. Δεν πρέπει απλώ να υπακούμε τυφλά στι αποφάσει του Συμβουλίου. Δεν μα εξέλεξαν γι' αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτε. Δεν είναι αυτό το καθήκον μα. Εμεί είμαστε το πιο δημοκρατικό θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκλεγχθήκαμε με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία από του Ευρωπαίου πολίτε. Επίσης μου είπατε ότι κανένας δεν έδωσε εξηγήσει ή κανένας δεν έκανε ελέγχους και ότι ε, επισύρονται εκατομμύρια προστήμων στις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω καθυστερήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει για την ε, ε ποινή να υπάρχει παράνομη ε, καθυστέρηση, ε, ζημία και σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ της καθυστέρησης και της ζημίας. Και σίγουρα κάποιες επιχειρήσεις ε, ίσως ε, ζημιωθούν από τις καθυστερήσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι για όλες τις καθυστερήσεις ευθύνεται το δικαστήριο ή για όλες τις καθυστερήσεις θα ενεργοποιηθούν πρόστιμα. Άλλωστε καθυστερήσεις έχουμε συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με λάθος επιχειρήματα προσπαθείτε να επιτύχετε το στόχο σας. Επίσης μερικοί μίλησαν και για μείωση του αριθμού των δικαστών. Ο κύριο Σβιέφκα είπε ότι εμεί ζητήσαμε μείωση του αριθμού των δικαστών. Λάθο. Εκτό κι αν ε, ε, δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι θα δούμε ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση. Γιατί δεν έχουμε μία απάντηση από το Γενικό Δικαστήριο. Γιατί δεν κάναμε ακρόαση με τους δικαστές ή με τον πρόεδρο του, Ευρω... του Γενικού Δικαστηρίου. Φαίνεται ότι μερικοί δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν τη γνώμη των δικαστών γιατί υπάρχουν κάποιες αλήθειες που τις, μας τις παρουσιάζουν μερικοί ως απόλυτες αλήθειες και θέσφατα, αλλά ίσως δεν ισχύει αυτό. Γιατί φοβάστε να ακούσουμε τους ίδιους τους δικαστές, τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Γιατί μερικές φορές σκέφτομαι, και ως βουλευτής αλλά και ως απλός πολίτης, αν το πρόβλημα βρίσκεται στο Γενικό Δικαστήριο, γιατί να μην ακούσουμε τον πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου και τους δικαστές. Γιατί έχω έγκυρες πληροφορίες ότι οι δικαστές ε, διαψεύδουν πολλά από τα θέματα που για μας είναι απόλυτες αλήθειες. Δεν ισχύει αυτό. Επίσης, εμείς αποφασίζουμε για μια διαδικασία. Αλλά και εμείς οι ίδιοι θα αξιολογηθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα κριθούμε για τις αποφάσεις μας. Επίσης, σας είπα ότι η συνθήκη της Νίκης και η συνθήκη της α, Λισαβόνας είναι υπέρ της α, σύστασης ειδικών δικαστηρίων. Και κατά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία διαπίστωσα ότι η ειδική η δικαιοσύνη, τα ειδικά δικαστήρια είναι τα καλύτερα. Γιατί οι ειδικέ δικαιοδοσίες με ειδικευμένους δικαστές κάνουν την καλύτερη δουλειά. Λόγω της σωστής, της ειδικευμένης κατάρτισης. Τώρα, με την κατάρτιση του ειδικού δικαστηρίου, ουσιαστικά αντιτασσόμαστε και καταστρατηγούμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και το μοναδικό ε, ειδικό δικαστήριο που έχουμε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας και που τώρα θέλουμε να καταργήσουμε, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να αυξήσουμε, να διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών στο γενικό δικαστήριο. Εγώ δεν συμφωνώ με τη γνώμη ενός συναδέλφου ότι στην αρχή είπαμε ναι στην αύξηση των δικαστών και τώρα λέμε όχι δεν ευσταθεί αυτό που μας είπατε. Ούτε είναι σωστός αυτός ο τρόπος να θέτε το θέμα. Εμείς είπαμε ναι στην αύξηση των δικαστών κατά 12 μόνο επιπλέον. Τώρα δεν λέμε όχι στην αύξηση των δικαστών, ε, όχι στο διπλασιασμό των δικαστών, στην αύξηση κατά 28 και στην κατάργηση ενό ειδικού δικαστηρίου που μέχρι στιγμής λειτουργήσε αποτελεσματικά και προς όλων των ενδιαφερομένων. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε με προκαταλήψεις, είτε είναι πολιτικές είτε είναι νομικές. Θεωρώ θα πρέπει να εγγύψουμε στο πρόβλημα με την δέουσα εντιμότητα. Την εντιμότητα που απαιτεί η σοβαρότητα του προβλήματος. Και να μην κολλάμε σε προκαταλήψεις. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό ε, προ την κυρία Χάουταλα και είπε από του 28 νέου δικαστέ οι 14 να είναι γυναίκε. Ναι, γιατί όχι. Μάλιστα, εγώ ήμουν πρόεδρο του Πορτογαλικού Δικηγορικού Συλλόγου και εφάρμοσα την ισότητα στον Δικηγορικό Σύλλογο τη Πορτογαλία. Και μάλιστα, ο Πορτογαλικό Δικηγορικό σύλλογο είναι ο μοναδικό δικηγόρικό σύλλογο στον κόσμο που η πλειοψηφία των γυναικών βρίσκονται σε ηγετικέ θέσει. Είναι ο μόνο δικηγορικό σύλλογο που έχει τόσες πολλέ γυναίκε στο προεδρείο του, στον κόσμο. Είμαι υπέρ τη ισότητα των γυναικών. Και υπέρ τη ισότητα όχι μόνο στο δικαστήριο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί όχι. Το θέμα είναι όμω, δικαιολογείται ο διπλασιασμό των δικαστών. Η αύξηση του κατά 28 επιπλέον. Σκεφτείτε το, κύριε συνάδελφε. Δικαιολογείται από τη μία η κατάργηση του δικαστηρίου δημόσιας διοίκηση και από την άλλη ο διπλασιασμό των δικαστών η αύξησή τους από 28 σε 56. Αυτά θα πρέπει να σκεφτούμε. Έτσι θα πρέπει να επιστρατεύσουμε εκατομμύρια κάθε χρόνο από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Ενώ ταυτόχρονα λέμε ότι κοπτόμαστε για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ζητούμε περικοπές. Συνέχεια μιλούμε για περικοπές δαπανών αν κάποιες δαπάνες είναι απαραίτητες, να τις κάνουμε. Αλλά πρώτα να δούμε αν είναι πραγματικά απαραίτητες. Αν δικαιολογούνται. Γιατί δεν μπορούμε να δεχόμαστε α, χωρίς έλεγχο κάτι που μας λέει και να μην το εξακριβώνουμε πρώτα, να μην το επαληθεύουμε. Νομίζω ότι ένα τμήμα της αλήθειας δεν έχει ακόμη ακουστεί και δεν έχει ακουστεί από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, από τους ίδιους τους δικαστές. Ποιος φοβάται να ακούσει τους ίδιους τους δικαστές. Γιατί. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με την πρότασή σας να... ή τέλος πάντων γενικότερα, το πω, πώς να προχωρήσουμε. Αυτό νομίζω θα το αποφασίσουν, θα το συζητήσουν μάλλον και θα το αποφασίσουν αύριο οι συντονιστές γιατί φαίνεται μάλλον περίπλοκο θέμα και χρειαζόμαστε κάποια συμφωνία μεταξύ των συντονιστών αν συμφωνείτε. Για την κυρία Χάουταλα έχω να πω ότι διαδίδονται πληροφορίες ότι κάποιοι περιμένουν τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Ο μέσος όρος για το 2014 ήταν 23,5 μήνες λιγότερο από δύο χρόνια. Επομένως αυτό είναι αντίθετο από το πρώτο που είπα. Ε, φαίνεται πως δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες, πάντως όχι σίγουρες. Η κυρία Ρέγνερ που δυστυχώς απεχώρησε μας είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα το νέο ίσως εσείς να γνωρίζετε καλύτερα από εμένα αλλά για μένα η πληροφορία ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν συμφωνεί με την προτινόμενη μεταρρύθμιση αυτό το στοιχείο για μένα είναι νέο και βέβαια είναι σημαντικό νέο ασφαλώς Α, ε, η κυρία Ντελβό επιθυμεί να επανέλθει. Κοιτάξτε, θέλω να υπενθυμίσω ότι το κείμενο δεν προβλέπει να δώσει γνώμη το δικαστήριο το άρθρο 281 λέει ότι ζητεί τη γνώμη του δικαστηρίου και γίνεται συζήτηση μεταξύ των μελών του δικαστηρίου. Έχουν υπάρξει και άλλες προτάσεις μεταξύ των δικαστών του πρωτοδικίου, αλλά τουλάχιστον στα επίσημα κείμενα δεν υπάρχει η επίσημη θέση του δικαστηρίου. Είναι υπόθεση που πρέπει να συζητήσουν οι δικαστές μεταξύ τους. Κάναμε μια επίσκεψη που εγώ θεωρώ ήταν επίσημη επίσκεψη στο Λουξεμβούργο συνήλθε και η Επιτροπή μας στο Λουξεμβούργο μαζί με τους δικαστές και του Γενικού Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου και η μόνη άποψη που ακούσαμε ήταν η άποψη του Προέδρου του Δικαστηρίου. Δεν μας ανέπτυξαν ενάντιες θέσεις ως θεσμικό όργανο, ερχόμαστε σε επαφή με θεσμικά όργανα. Τώρα αν υπάρχουν εντός του οργάνου δικαστήριο αποκλίνουσες απόψεις, κοιτάξτε αυτό είναι άλλη υπόθεση, αλλά και εδώ στο κοινοβούλιο υπάρχουν διαστάσεις απόψεων, αλλά τελικώς καταλήγουμε σε μία απόφαση. Σύντομα παρακαλώ κύριε. Αγαπητή κύριε Τελφό, είναι προφανές ότι η επίσημη θέση και η πρωτοβουλία προήλθαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά επειδή η κατάσταση είναι περίπλοκη, αξίζει να ακούσουμε τους ίδιους τους δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου. Γιατί εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Στο Γενικό Δικαστήριο είναι το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Στους δικαστές και στους υπαλλήλους. Γιατί να μην τους ακούσουμε. Με προβληματίζει και με ανησυχεί γιατί ασκείται αυτή η πίεση να μην έχουμε ακρόση με τους δικαστές που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι για να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί να μην τους ακούσουμε, να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από τις παρεμβάσεις τους, να τις σταθμίσουμε, να τις αξιολογήσουμε και να λάβουμε τεκμηριωμένα την απόφασή μας. Τώρα, να αποκλείουμε εξ αρχής οποιαδήποτε ακρόαση με τον πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου και με τους δικαστές, τι να σας πω, με προβληματίζει και με ανησυχεί το μάλα. Είναι αδιανόητο το Κοινοβούλιο να αρνείται να ακούσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους για το πρόβλημα, του δικαστές του Γενικού Δικαστήριου, στο οποίο και εντοπίζεται το βασικό πρόβλημα. Ε, okay. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να συναντηθείτε με τους κοιόδης συγητές στο Στρασβούργο στις 28 Τετάρτου. Σι λέει ο συγητής. Δηλαδή ναι. Και αν δεν γίνεται στο Στρασβούργο, πολύ ευχαρίστω στις Βρυξέλλες, ε, αν γίνεται κύριε Πρόεδρε. Well, the proposal is to, to hold the... Κοιτάξτε, η πρόταση είναι να γίνει η συνάντηση 28 Τετάρτου, 28 Απριλίου, δηλαδή Στρασβούργο. Καταρχάς, ναι. Θα φροντίσω να κανονίσω το πρόγραμμά μου για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτή τη συνεδρίαση. Okay. So, ε, Πρόεδρος. Εντάξει, αυτό λοιπόν θα είναι το επόμενο βήμα και θα μπορέσει, θα μπορέσει να συζητηθεί το θέμα αυτό μεταξύ των συντονιστών. Αν δεν υπάρχουν άλλες επιθυμίες να λάβετε το λόγο, να προχωρήσουμε τότε στο υπαριθμό 6. Εξέταση της εκθέσεως για την προστασία της τεχνογνωσίας και δίνω το λόγο στην κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φτάνουμε σήμερα στην τρίτη μας ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση οδηγίας για την προστασία της τεχνογνωσίας και των εμπιστευτικών πληροφοριών. Έχω ήδη καταθέσει το σχέδιο εκθέσεώς μου στη Γραμματεία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις 10 Φεβρουαρίου. Όλες οι μεταφράσεις είναι διαθέσιμες εδώ και τρεις εβδομάδες περίπου. Αν λοιπόν είχατε την διάθεση, είχατε και την ευκαιρία να τις εξετάσετε και έτσι θα σας αναπτύξω λίγο τις βασικές κατευθύνσεις. Τα έχω πει ήδη, αλλά το επαναλαμβάνω ότι δέχθηκα ευνοϊκά το σχέδιο οδηγίας που είναι αποτέλεσμα των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που θεωρώ ότι είναι χρήσιμη ως βάση εργασίας και προσεπάθησα να βελτιώσω, να εμπλουτίσω, να καταστήσω ακριβέστερο, παρά να ανατρέψω την ισορροπία και να αλλάξω τον τελικό σκοπό που είναι η προστασία της τεχνογνωσίας, δηλαδή να δοθούν τα όπλα στις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αμήνονται κατά της παράνομης διάδοσης εμπιστευτικών πληροφοριών για την τεχνογνωσία τους. Άρα προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινή νομική βάση, μια κοινή έννοια σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό απόρριτο, μια τέτοια λοιπόν κοινή αντίληψη που θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ασφάλεια των επιχειρήσεων στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των η ανταλλαγή προφοριών είναι απόλυτα ζωτική και κρίσιμη, αναγκαία, για να διευκολυνθεί η προώθηση, η ανάπτυξη της ε, βιομηχανίας της γνώσης, που είναι και το σήμα κατά τεθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν κλίμα εμπιστοσύνης για να αναπτυχθούν οι ε, ανταλλαγές αυτές τεχνογνωσίας και που χρειάζεται ε, ρύθμιση το πεδίο αρμοδιοτήτων είναι το εξής. Προτείνονται αστικού χαρακτήρα μέτρα για την αντιμετώπιση των παράνομων διαδόσεων του βιομηχανικού απορρίτου, διότι αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει και τα όρια της ευθύνης εκείνων που χρησιμοποιούν ενδεχόμενα παράνομα μέσα για να αποκτήσουν τις σχετικές πληροφορίες. Άρα δεν πρόκειται, καθόλου μάλιστα, για οποιαδήποτε άρση της υποχρέωσης διαφάνειας, για παράδειγμα, από, για τα έγγραφα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Το ίδιο, οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στις δημόσιες αρχές οφείλουν να προστατεύονται σε ό,τι αφορά την κατοπινή χρήση τους. Αν δηλαδή μια επιχείρηση υποβάλει μια προσφορά για μια δημόσια προμήθεια στην οποία περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες στο περί της στρατηγικής της αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να αναμένει από τις δημόσιες αρχές ότι αυτές θα σεβαστούν την ευθύνη που φέρουν, την νομική ευθύνη που φέρουν όσον αφορά την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Ωστόσο, το επαναλαμβάνω ρητά, στην ε, τροπολογία μου παριθμών 5. Αυτή η υποχρέωση τήρηση τη εμπιστευτικότητας για τι δημόσιε αρχέ καλύπτεται και από την παράγραφο 3 του άρθρου 3. Προσπαθώ επίση να άρω κάποια, κάποια κενά στο κείμενο, στα άρθρα 2, 3 και 4, που είναι εκείνα που προβλέπουν τον ορισμό του βιομηχανικού απορρίτου και τη ε, χρήση του, για τη χρήση του. Και προβλέπω και μια ε, προθεσμία προσφυγής της τάξης των τριών ετών. Η προθεσμία που βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι το λιγότερο ενός έτους και το πολύ δύο ετών μου φαίνεται ανεπαρκή. Γι' αυτό προβλέπω εγώ τρία έτη που θα επιτρέπουν στον προσφεύγοντα να ε, φτιάξει, να, στερεώσει την υπόθεση καλύτερα δηλαδή, εφόσον πρόκειται ενδεχόμενα για ένα θέμα ε, περίπλοκο το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στις ε, δικαστικές αρχές και να είναι επομένω γερά τεκμηριωμένο και θεμελιωμένο. Άρα προθεσμία προσφυγή των τριών ετών ως ε, απαραίτητο στοιχείο αυτής της κοινή προσέγγισης για να αποφευθεί και η άγρα δικαστήριο, το forum shopping. Η διάταξη λοιπόν βασίζεται στο δίκαιο αστικό και εμπορικό της κάθε χώρας μέλους. Περί αυτού πρόκειται. είναι. Αυτό είναι το πεδίο αρμοδιοτήτων όπου τοποθετούμεθα. Άρα αστικό και εμπορικό δίκαιο της κάθε χώρας μέλους. Εκεί καθορίζονται οι παράνομες πράξεις. Προβλέπω και μια ενίσχυση της θέσης της επιχειρήσεως στον αγώνα της κατά των ε, παράνομων μεθόδων έτσι ώστε ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 4 να αποφευθεί λοιπόν ότι αυτές οι εξαιρέσεις θα χρησιμοποιηθούν ως προπέτασμα για εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε πρακτικές αντίθετες με τα ε, ήθη των, ε, τα συναλλακτικά ήθη. Επίσης, θέλω να επαναλάβω σαφώς ότι το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, κατά την άποψή μου, δεν παραβιάζει τις ελευθερίες. Θέλω να διατηρηθεί δηλαδή η εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή στο άρθρο 4. Αναφέρομαι ειδικά στην, στον σεβασμό της ελευθερίας πληροφόρησης. Έχω λοιπόν εμπλουτίσει το αρχικό άρθρο 4, προσθέτοντας κάποιες διευκρινήσεις και βάζω και κάποιες συγκεκριμένες ρητές αιτιολογικές σκέψεις ότι η ζωτικότητα της κοινωνίας, έχει σχέση βεβαίω και με την ελευθερία του τύπου κτλ. Ε, σε καμιά περίπτωση λοιπόν το κείμενο αυτό δεν θα επιτρέπει να προσβληθεί το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Και κανείς δεν θα μπορεί να δεχθεί την μομφή ότι χρησιμοποίησε με θεμητό τρόπο την ελευθερία ενημέρωσης Ακόμα και αν έγινε αυτό στη βάση κάποιων εγγράφων που ενδεχομένως να περιλαμβάνουν και εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες. Διευκρινίζω ακόμα στην τροπολογία μου 7 την ανάγκη προστασίας των πηγών. Μου φαίνεται επίσης σημαντικό οι ε, ρήτρες του άρθρου 4 στο κείμενο της οδηγίας που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκταθούν και σε ενδεχόμενα ποινικά μέτρα, μέτρα ποινικού χαρακτήρα που μπορούν να ληφθούν από τις χώρες μέλη όταν θα έρθουν όταν θα φτάσουν δηλαδή στη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Δηλαδή μπορούν να βγουν παραπέρα, οι χώρες μέλη να προχωρήσουν παραπέρα και να υιοθετήσουν και μέτρα ποινική προστασία της ε, προστασία των επιχειρήσεων. Αυτό βεβαίω είναι ένα κάτω δικαίου που δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, το ποινικό δηλαδή. Εκεί πρέπει να προβλεφθεί μηχανισμό που να αντιγράφει τα όσα έχουμε κάνει παλαιότερα για τη μεταφορά στα εθνικά δίκαια της οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών. Έχω βάλει λοιπόν όπως είπα στο άρθρο 4 τις ε, εγγύσεις αυτές διότι έχουμε ακούσει ανησυχίες να διατυπώνονται από ορισμένους τομείς της κοινωνίας των πολιτών, από ορισμένες ενώσεις σε κάποια μέσα ε, ενημέρωσης. Αυτά βεβαίως πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και έχω την ευήκον ους σε αυτά. Θα ήθελα επίσης να παρασχεθεί αποτελεσματική προστασία σε δίκαιη στην αρχή της δίκαιης δίκης και στην κατατιμωλία παράσταση. Στο άρθρο 8 που είχε προταθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το άθρο λοιπόν μου φαινόταν υπερβολικό όσον αφορά την προστασία του εμπορικού απορρίτου. Έχω λοιπόν καταθέσει τροπολογίες 31, 32 και 33 που εγγυώνται ότι οι διάδικοι θα έχουν ελάχιστη εγγυημένη πρόσβαση στο σύνολο των ε, ακροαματικών διαδικασιών και των εγγράφων. Για να είναι εγγυημένη λοιπόν η δίκαιη δίκη. Η διαδικαστική πτυχή αναφέρεται σε υποθέσεις που έχουν σχέση με την χρήση, διάδοση και ούτω καθεξής κατά παράνομο, κατά παράνομο τρόπο πληροφοριών ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα, Βεβαίω οι χώρε μέλη μπορούν να προχωρήσουν και περισσότερο στην νομοθεσία που θα θεσπίσουν. Σεβόμενες βέβαια πάντα την ανάγκη ε, εγγύησης της αρχής της δίκης δίκης. Ε, για να μην μακρηγορώ κύριε Πρόεδρε, αυτές είναι οι πιο βασικές τροποποιήσεις καθώς και προσθήκες που έχω που υποβάλλω μάλλον στην ε, νομική επιτροπή σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εντάχει και μετά έχω και ένα τελευταίο που ακόμα δεν έχω περιλάβει στο σχέδιο εκθεσεώς μου αλλά που ε, αναγνωρίζω ότι έχει σημασία τώρα για το χρονοδιάγραμμα όπως έλεγα Έχει δημοσιευθεί το σχέδιο εκθέσεώς μου εδώ και αρκετές εβδομάδες όπως εξήγησα στην αρχή της ομιλίας μου. Επομένως η προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών λίγη στις 26 Μαρτίου. Μπορεί να γίνει μια νέα συνάντηση της Επιτροπής μας για να συζητηθούν οι τροπολογίες περί τα μέσα Απριλίου και ίσως μετά θα μπορούμε να ψηφίσουμε στη διάρκεια της συνεδριάσεως του Μαΐου. Πριν να τελειώσω, ένα τελευταίο θέμα κύριε Πρόεδρε, αν με επιτρέπετε. για τα θέματα που είχαν τεθεί και στη δημόσια διαβούλευση που είχε οργανώσει η Επιτροπή στις 20 ε, Ιανουαρίου για την ε, κινητικότητα των επαγγελματιών δεν θέλω εγώ από μόνη μου να περιλάβω τροπολογίες, προτάσεις, τροποποιήσεις για το θέμα αυτό της επαγγελματικής κινητικότητας στο σχέδιό μου αφενός διότι θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κοινό θεμέλιο για την προστασία του εμπορικού απορρίτου κτλ. θα συμβάλλει στην κινητικότητα αυτή, αλλά και διότι οι άλλες πολιτικές ομάδες είναι αρκετά γόνιμες σε αυτό το θέμα. Νομίζω μόνο ότι ένας αριθμός εγγύσεων υπάρχουν έτσι ώστε αυτό το κοινό θεμέλιο για την προστασία του εμπορικού απορρίτου να μην αποτελέσει εμπόδιο στην κινητικότητα των επαγγελματιών. Υπάρχουν άλλωστε επιχειρήματα που ε, μπορώ να προβάλλω ε, στις απαντήσεις που ε, ενδέχεται να κληθώ να δώσω σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Και τέλος, προστασία της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας, που είναι και ο όρος κλειδί για την πρόοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες είναι και το απαραίτητο καύσιμο σε αυτή την οικονομία της γνώσης που τόσο χρειαζόμαστε. Επομένως πρέπει να εργαστούμε επί τη διατήρηση της ισορροπίας αυτής για να μπορούν να κυκλοφορούν, να συνεχίσουν να κυκλοφορούν οι πληροφορίες μέσα στον ευρωπαϊκό μας χώρο. Αναμένω με αληθινή ανυπομονησία τις τοποθετήσεις των συναδέλφων μου. ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με παραγωγικό τρόπο με συνεργασία των σκιωδών εισηγητών αλλά και των υπολείπων συναδέλφων που ενδιαφέρονται. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών που λήγει το μεσημέρι στις 26 Μαρτίου. ήθιστε στην Επιτροπή μας να καθυστερούμε δυστυχώς. Γι' αυτό ακριβώς επειδή έχουμε μείνει πίσω και σήμερα να σας ζητήσω να είστε λακωνικοί στα σχολεία σας. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, για την εργασία που ε, έκανε ε, υπογράφοντας και κάποια, ε, ε, υπογραμμίζοντας και κάποια στοιχεία τα οποία είναι καινούρια. Θα ήθελα όμως να κάνω και δύο παρατηρήσεις. Μία γενικού χαρακτήρα και το λέω και υπό το φως της συζήτηση στην οποία έλαβα μέρος σε άλλες επιτροπές, ιδιαίτερα δε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Το κείμενο της Κομισιόν όσον αφορά το βιομηχανικό αφόρητο φαίνεται, μπορεί μάλλον να εμφανιστεί σαν ένα ε, κείμενο καθαρής συντήρησης, ενώ εμείς θέλουμε να διευρύνουμε ε, το θέμα αυτό όχι μόνο υπέρ των επιχειρήσεων που υφίστανται ήδη, αλλά και ε, για να ρυθμίσουμε μία αγορά η οποία μπορεί και να διευρυνθεί και να ανοίξει. Επομένως, να μην μπερδεύουμε την προστασία με την αυτάρκεια να κάνουμε αντιθέτως τη λέξη αυτή ε, συνώνυμη με την πραγματική ανταγωνιστικότητα ή τον πραγματικό ανταγωνισμό. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα ευαίσθητα. Το πιο ευαίσθητο είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με, του, με την εργασία των ανθρώπων, ιδίω σε υψηλότερο επίπεδο, εκεί όπου η καινοτομία είναι ακριβώς η βάση της εργασίας τους. Εάν εμείς προστατέψουμε αυτούς τους επαγγελματίες, όχι μόνο τους απαγορεύουμε κατά κάποιο τρόπο, ζημιώνουμε την δυνατότητα που έχουν να κάνουν προτάσεις στην αγορά εργασίας που τους αφορά, αλλά ε, κατά κάποιο τρόπο δημιουργούμε πρόβλημα και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Εάν δεν αναγνωριστεί η, ε, αξία της δημιουργίας, χωρίς να το θέλουμε, στην ουσία ζημιώνουμε και το άτομο και την επιχείρηση στην οποία το άτομο αυτό είναι εμπλεγμένο και επομένως, και επομένως ε, κυρίως ζημιώνουμε αυτήν την πνευματική τους εργασία, την διαδικασία της σύλληψης της ιδέας, του σχεδιασμού ε, και χάνουμε την ευκαιρία να διευθετήσουμε αυτές τις ιδέες με καινοτόμο τρόπο έτσι ώστε να αποκτήσουμε να πραγματική αξία ε, αυτό που οι άνθρωποι αυτοί κάνουν. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Ε, ε, πνευματική παραγωγή φυσικά αλλά που τελικά φτάνει στην πραγματική παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή, ε, παραγωγή και παροχή υπηρεσιών κτλ. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να μας απασχολήσει και όσον αφορά τις δράσεις της δημόσιας διοίκησης που συχνά κρύβονται πίσω από το απόρριτο έτσι ώστε να έχουν ε, στην διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, ε, δραστηριοτήτων τους κάποια διακριτικά περιθώρια πολύ μεγάλα και πολύ ύποπτα. Αναφερόμαστε εδώ στη σχέση με ένα σύστημα το οποίο τίνει να είναι ανοιχτό ε, σε εξωτερικές συνθήκες και προϋποθέσεις σαν αυτές που εσείς αναφέρατε προηγουμένως όσον αφορά τους διαγωνισμούς και τις προμήθειες, κυρίως δε τους μεγάλους δημόσιους διαγωνισμούς. Πρόκειται για πολύ ευαίσθητα θέματα λοιπόν, τα οποία ε, θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν ε, με πολύ σωστό τρόπο. Η υποβολή των τροπολογιών φαντάζομαι ότι θα μας δώσουν την δυνατότητα να βρούμε θετικές λύσεις σε αυτά τα δύο σημαντικά θέματα. Υπάρχει κι άλλο ένα, η παραγραφή και ο χρόνος παραγραφής. Εγώ θεωρώ ότι είναι και αυτό ευαίσθητο θέμα. Προφανώς η επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής ε, δίνει δυνατότητα προσφυγής. Ε, αυτό εκ πρώτης όψεως, γιατί στην ουσία δεν είναι έτσι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί, γιατί και γι' αυτό ακριβώς θεωρούσα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη την πρόταση της Κομισιόνα, ε, ο, αυτός ο μακρύτερος χρόνος δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα γνώσης στον εφεσιβάλλοντα, αλλά παρόλα αυτά στην ουσία μειώνει την, ε, το έβρος και τη σημασία της ε, παράνομης πράξης. Ε, ε, γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει κοντινά χρονικά να βρισκόμαστε στην, στις διαδικασίες. Γι' αυτό συμφωνούσαμε με το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος, υποτίθεται ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια αναπαράσταση ας πούμε των περιστατικών με πιο πλήρη τρόπο, αλλά παρόλα αυτά όσο περνάει ο καιρός αλλάζουν και οι συνθήκες της αγοράς αγοράς και επομένως αλλοιώνεται και η φυστάμενη ζημία. Νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο να προσανατολιστούμε προς ε, την, πρόταση της, την αρχή πρόταση της Κομισιόν και να μην λάβουμε υπόψη μας στο Συμβούλιο το οποίο προσπαθεί να αλλάξει τη φύση του πράγματος ε, και μετά τροποποιεί στην ουσία την πραγματική αξία που θα πρέπει ουσιαστικά να αναγνωριστεί και επομένως να πληρωθεί σαν τέτοιο. Ευχαριστώ. Yeah, very much. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ρέγνερ. First of all, I'd like to thank the... Ευχαριστώ καταρχήν την εισηγήτρια. Συμφωνώ ότι για τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να προσπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αλλά συμφωνώ και με τον κύριο Κοφεράτη ότι δεν συμμεριζόμαστε με τη γενικά θετική αξιολόγηση του σχεδίου οδηγίας γιατί δεδομένου του εφνομοθετήν και επειδή ήδη έχουμε προστασία των εμπορικών απορρίτων σε εθνικό επίπεδο, μια οδηγία θα πρέπει να σημαίνει εξασφάλιση ε, της ασφάλειας δικαίου για όλους τους ενδιαφερομένους. Και έχω και συγκεκριμένου προβληματισμούς, ε, γι' αυτό και θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Για παράδειγμα, στο θέμα των ορισμών. Ποιες είναι οι πληροφορίες που τη χάνουν προστασίας δεν μιλούμε για καινοτόμε πληροφορίες ε, επιχειρηματικές. Δεν επικεντρωνόμαστε στο είδο των πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται και δεν αποκαλύπτονται ακριβώς επειδή έχουν ένα καινοτόμο δυναμικό. Ούτε αποκλείονται οι πληροφορίες που οφείλουν να, να αποκαλύπτουν για κανονιστικούς λόγους οι επιχειρήσεις. Σε κράτη-μέλη είχαμε περιπτώσει όπου κυβερνήσει δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα ελευθερίας πληροφορίας γιατί αυτό θα σήμαινε αποκάλυψη ε, εμπιστευτικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Αυτό όμως είναι κάπως προβληματικό όταν μιλούμε για την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να διατηρούν τους ειδικότερους ορισμούς τους αυτού που ισχύουν στι εσωτερικέ του νομοθεσίε. Τώρα, το ίδιο ισχύει και για τον κατάλογο των εξαιρέσεων και των περιορισμών. Δεν αναφέρεται το σαφέ δημόσιο συμφέρον ή εξαιρέσει λόγω δημόσια υγείας ή περιβάλλοντο. γιατί αποκάλυψη περιφερειών που είναι προ όφελο του γενικού συμφέροντο από κάποιου πληροφοριοδότε ή καταγγέλλοντε, ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αθέμητη αποκάλυψη εμπορικού απορρίτου Επίσης, το θέμα της νομοποίησης για την άσκηση της ελευθερίας της πληροφορίας ή της ελευθερίας έκφρασης. Τέτοια θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά ανεφόρων, χωρίς επιβέρους χαρακτηρισμούς. Επίσης, δεν προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματα των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους στον κατάλογο με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς. Και από αυτή την άποψη Φοβόμαστε ότι ίσως η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής παγώσει κάπως την ε, κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό θα καταθέσουμε τροπολογίες για να βελτιώσουμε τα σχετικά εδάφια. Για παράδειγμα, το, τη συγκεκριμένη προθεσμία οριοθέτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Κοφεράτη ότι σω θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν έχουμε όμω αγωγέ ει βάρο πρώην εργαζομένων, η ανώτατη περίοδο ε, θα πρέπει να είναι ένα έτος. Επίση, θα προβλέπουν κάποιε αποζημιώσει για κάποιου που έχουν κατα... κατηγορηθεί ε, εσφαλμένα ότι έχουν αποκαλύψει εμπορικό, εμπόριτο, ε, αυτό έχει θίξει την ε, αξιοπρέπεια του επιθύμητους, ειδικά για τις μικρομέσες επιχειρήσεις. Γιατί μπορεί μεγάλε εταιρείε να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να κρατήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μακριά από την αγορά και να. Ε, επειδή ακριβώ έχουν πολύ περισσότερους πόρους και μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια. Τέλος, για τη διατύπωση που χρησιμοποιεί, την ορολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν συμφωνώ με τον όρο ε, παραβίαση αντί για ε, παράνομη ή αθέμητη αποκάλυψη για την επιβολή κυρώσεων, γιατί στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει το εμπορικό απόρριτο δεν εμπίπτει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκεί χρησιμοποιείται επιβολή κυρώσεων στο διαδικασία ε, επί παραβάση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι το εμπορικό απόρριτο δεν πρόκειται να αποτελέσει τμήμα των δικαιωμάτων πνευματικής διαδικασίας. Τότε γιατί χρησιμοποιείται στο TTIP το εμπορικό απόρριτο στο κεφάλαιο με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης χρησιμοποιούν το εμπορικό απόρριτο στα πλαίσια των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες μέλη. Άλλες φορές εμπίπτει στο δίκαιο ανταγωνισμού. δημιουργεί σύγχυση το ότι συμπεριλαμβάνει το εμπορικό απόρριτο στα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία στην Διαδηλαντική Συμφωνία TTIP. Και αμφιβάλλω για το κατά πόσο είναι σωστή η νομική βάση που χρησιμοποιεί η οδηγία για την υποβολή αυτή τη πρόταση. Όλε αυτέ τι διευκρινήσει θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ε, ρόλο των εμπορικών απορρίτων στις διαπραγματεύσεις TTIP. Ο κύριος Ράνεφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λεγκρίπ για την εξαίρετη εργασία της. Συμφωνώ με τη θέση που έχει λάβει, δηλαδή ότι δεν είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί πλήρως ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, επιβάλλονται ε, τροποποιήσεις, αλλαγές οι οποίες θα βελτιώνουν το τελικό κείμενο στηρίζω την θέση της κυρίας Λεγκρίπε να γίνει πιο συγκεκριμένη η έννοια του εμπορικού ε, απορρίτου. Επίσης, ότι ε, συμφωνώ μαζί της ε, ότι θα πρέπει να προστατεύονται και όλα τα στοιχεία τα οποία ε, ε, σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης. Συχνά είναι δύσκολο να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει εμπορικό απόρριτο. Νομίζω ότι θα πρέπει οι ίδιες οι επιχειρήσεις να ορίζουν τι ακριβώς αποτελεί για αυτούς ε, απόρριτο. Επίσης, ε, η εναρμόνιση ε, των κανόνων όσον αφορά τον χρόνο προσφυγής είναι κάτι μεγάλης σημασίας και θα πρέπει ομοιογενώς να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι τα τρία χρόνια είναι αρκετά γιατί ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προτείνουν ε, μεγαλύτερο διάστημα για μεγαλύτερη προστασία και αυτή ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο ανάμεσα στα τρία και τα 6 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μαρίνου Πίντου. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητριά μας Φαίνεται από την παρουσίαση ότι είναι πολύ άρτιο το έργο της. Έχω βέβαια κάποιες επιφυλάξεις και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για επιμέρους σημεία. Έχουμε σήμερα κάποιους που είναι επιφορτισμένοι με την προάσπιση των απορρίτων, αλλά έχουμε και άλλους που το καθήκον τους ή μάλλον το έργο τους είναι να παραβιάζουν και να αποκαλύπτουν απόρριτα. Η λογική του απορρίτου ε, προϋποθέτει την απόκρυψη από την κοινωνία κάποιων ε, ζωτικών πληροφοριών που επηρεάζει την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό και έχουμε ε, τη λειτουργία των δημοσιογράφων που η βασική τους αποστολή είναι να παραβιάζουν απόρριτα. Τώρα να ποινικοποιούμε ή την παραβίαση του εμπορικού απορρίτου ή να προστατεύουμε υπερβολικά το εμπορικό απόρριτο, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο. Γιατί κινητοποιούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και κινητοποιούμε το νομικό μας οπλοστάσιο για να προστατεύσουμε μερικές φορές σε κάποια θέματα που είναι ιδιωτικά συμφέροντα ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε ως απόρριτο κάθε πληροφορία που η αποκάλυψη της δεν επηρεάζει ή δεν θίγει ε, σοβαρά τα ένομα συμφέροντα μιας επιχείρησης. Είναι προφανές ότι η ίδια η επιχείρηση θέλει να κρατήσει μυστικές κάποιες πληροφορίες, ε, να μην φτάσουν στην κοινή γνώμη για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά το δημόσιο συμφέρον προϋποθέτει ή απαιτεί την γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών. Γι' αυτό και θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη σημασία της ε, δημοσιογραφικής λειτουργίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να ορίσουμε καλύτερα την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, γιατί για να προστατεύσουμε απόρριτα θα πρέπει να το κάνουμε στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος ακόμη και αν αυτό το δημόσιο συμφέρον απορρέει από μια ιδιωτική δραστηριότητα. Αλλά θα πρέπει να ορίσουμε σωστά την έννοια του δημοσίου συμφέροντο. Μόνο τότε είναι θεμητό να απαγορεύσουμε ή να επιβάλλουμε κυρώσει για την παραβίαση του απορρίτου. Μόνο όταν δικαιολογείται από λόγου δημοσίου συμφέροντος. Φυσικά με πλήρη σεβασμό του ελεύθερου τύπου και τη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων. Γιατί πολλέ φορέ, επαναλαμβάνω, το έργο των δημοσιογράφων η η παραβίαση των απορρίτων που θα ήθελα να είναι πιο καλά προστατευμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαν Ζαβά, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Λεγκρίπ και τη συγχαίρει θερμά γιατί συνεχίζει την ισορροπημένη προσέγγιση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εισηγήτρια υπέβαλε οκτώ διαφορετικούς τομείς. Εγώ θα σταθώ σε έναν μόνο, όπου έχουμε πρόβλημα με τις τροπολογίες 4 και 17. Θεωρούμε ότι οι τροπολογίες αυτές περιορίσουν την Γενική Αρχή της Ελευθερίας, της ε, ανεξάρτητης δημιουργίας και της ε, καινοτόμας μηχανικής. Γιατί αυτές οι αρχές που έχουν εξεταστεί διεξοδικά είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας πραγματικά ανταγωνιστικής ε, εσωτερικής αγοράς και την προώθηση της καινοτομίας. Χρειαζόμαστε αυτή την ανταγωνιστικότητα ε, και τον ανταγωνισμό στην καινοτομία. Και μάλιστα κάποια προϊόντα που δεν ε, τυχάνουν προστασία από τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία και αποκτώνται με έντιμα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελεύθερα και από άλλου προ όφελο τη οικονομική ε, επίδοση ε, του συνόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προ το συμφέρον των καταναλωτών τη. Κατά τη γνώμη, οι τροπολογίε αυτέ ίσω δημιουργήσουν νέου φραγμού στη χρήση πληροφοριών και γνώσεων που λαμβάνονται με έντιμα μέσα, χωρίς να παραβιάζεται κανένα, κανένας νόμος ή καμία σύμβαση. Βέβαια, κυρία Λεγκρίπ ε, έθεσε το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού. Η τροπολογία 17 τροποποιεί το άρθρο 4 και χαρακτηρίζει αθέμητη την απόκτηση ενός εμπορικού απορρίτου που θα μπορούσε να είχε ε, ληφθεί με έντιμα μέσα και χωρίς παραβίαση σύμβασης αν αυτή η απόκτηση εξυπηρετεί σκοπό που θεωρείται αντίθετος σε έντυμα συναλλακτικά ήθη. Και τονίζω αυτό το εξυπηρετεί το σκοπό, γιατί αν υπάρχει αδικοπραξία, αυτό αυτή δεν αφορά την ίδια την απόκτηση, που είναι το αντικείμενο της οδηγίας, αλλά την, ε, ε, στην ακόλουθη συμπεριφορά του αποκτήσαντος. Οπότε δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Και μας προβληματίζει η τροπολογία 17 για το λόγο αυτό. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι υπάρχει και ένα τελείως διαφορετικό θέμα που φαίνεται να καλύπτουν οι τροπολογίες και που πάλι εκπίπτουν το πεδίου εφαρμογής οδηγίες. Ε, γιατί μιλούν για θέμητο ανταγωνισμό, για εσφαλμένες διατυπώσεις, για σύγχυση της αγοράς ή παραπλάνηση των καταναλωτών. Τέτοιες συμπεριφορές εμπίπτουν στους κανόνες για τον αθέμητο ανταγωνισμό και μπορεί να μην υπάρχει ως εναρμόνιση, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο της συγκεκριμένης οδηγίας. Είναι το μόνο πρόβλημα πάντως που έχουμε με τις τροπολογίες της ε, κυρίας Λεγκρίπ. Γενικώ ε, χαιρετίζουμε τις προτάσεις της και συμφωνούμε μαζί της γιατί θεωρούμε ότι βελτίωσε την ισορροπία του κειμένου. Σε τη φορά τα σχόλια των ε, λοιπόν Ευρωβουλευτών, θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι η οδηγία δεν αναφέρεται σε ισχύοντες κανόνες ε, που διέπουν την αποκάλυψη πληροφοριών στις δημόσιες αρχές και λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δεν προβλέπει όρια ή δεν τροποποιεί την πρόσβαση ε, πολιτών ή οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών για θέματα που φορούν την υγεία, το περιβάλλον ή συναφείς πληροφορίες. Τέτοια θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ε, καλύπτονται από τον κανονισμό 1049 και η προστασία του εμπορικού απορρίτου ισχύει εδώ και πολλά χρόνια στα κράτη-μέλη. Αυτό που επιδιώκουμε με την πρότασή μα είναι να την εναρμονίσουμε, να την αποσαφηνίσουμε και να προβλέψουμε κατάλληλου περιορισμού και ασφαλιστικέ δικλείδε. Και σε καμία περίπτωση δεν αυξάνουμε την προστασία του εμπορικού απορρίτου. Η εντολή μα είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερη εναρμόνιση και να βελτιώσουμε τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και τις καινοτομίες με προνομιακούς εταίρους. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένη πρότασης. Και από αυτήν την άποψη θεωρούμε ότι οι ασφαλιστικές δικλείδες που τις αναγνωρίζουμε ε, ως θεμελιώδους σημασίας και ακριβώς έτσι με το κείμενο αυτό διευκρινίζονται και για την ελευθερία έκφρασης ε, ισχύει αυτό που είπε η κυρία Βίπερς που θα καταθέσει και τροπολογίες. Τέλος. Το θέμα της αλληλεπίδρασης του εμπορικού απορρίτου με την επαγγελματική κινητικότητα. Δεν πιστεύουμε ότι η πρότασή μας θα επηρεάσει αυτή την επαγγελματική κινητικότητα. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορούν ελεύθερα να αλλάζουν δουλειά. Βέβαια, οι πληροφορίε που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην νέα θέση είναι αυτέ που ήδη με βάση του ισχύοντε κανόνε απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν. Γιατί κάτι τέτοιο θα, μπορούσαν, θα μπορούσε να επηρεάσει ε, τα συμφέροντα του προηγούμενου εργοδότη. Θεωρούμε ότι υπάρχει βέβαια τέτοια δυνατότητα και αναφέρεται και στη μελέτη επιπτώσεων μας ότι με την ε, εξασφάλιση μεγαλύτερη ενάρκεια και σαφήνειας θα βελτιωθεί η επαγγελματική κινητικότητα και θα μειωθεί η εξάρτηση από ρήτρε ε, μη ανταγωνισμού που ισχύουν σε μερικού τομεί. Οπότε, επαναλαμβάνω, επικροτούμε το σχέδιο έκθεση τη συγκήτρια, χαιρετίζουμε το έργο τη Επιτροπή και περιμένουμε με δημονία τις υπόλοιπες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you very much, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σέντερ. Θα ήθελα απλώς να κάνω μια ερώτηση αν θέλει να σχολιάσει σχετικά με τη διαδικασία TTIP, διαπραγματεύσεις TTIP. Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα ε, θέσατε δύο ε, ερωτήσεις. Ε, γιατί χρησιμοποιούμε την λέξη παραβίαση, γιατί είναι μια γενική ε, ε, λέξη την οποία δεν χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα ε, στο κείμενο αυτό. Όσον αφορά το TTIP πρέπει να σας πω ότι και στην ΤΡίψε υπήρχε η κάλυψη και προβλέποντο ούτως ή άλλως οι διμερείς συμφωνίες στα πλαίσια της ΤΡίψε Είπα και προηγουμένως και το έχω ξαναπεί και στην Επιτροπή εδώ ότι σαφώς δεν έχουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο σε αυτό την, σε αυτό το θέμα θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει με την πρόταση αυτή, τι θα αποφασίσουν μάλλον οι συνομοθέτες ε, και επομένως ε, δεν θα συζητηθεί κάτι τέτοιο μέχρι ότου στο καταστατικό προβλεφθεί κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λεγκρίπ θέλει να απαντήσει. Όχι. Εντάξει. If uh, Επομένως μπορούμε να, ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να, να συνεχίσουμε με το σημείο 7 σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά τη συμφωνία TTIP και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Βόσα, αλλά πριν του δώσω το λόγο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ε, από τη στιγμή που η ψηφοφορία ε, για την γνωμοδότηση αυτή έχει προβλεφθεί για τη 16η Απριλίου η ε, εκπνοή των τροπολογιών θα είναι στις 26 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα, ημέρα Πέμπτη. Κύριε Βός, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, <clears throat> ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα για την ίδια τη γνωμοδότηση που ασχολείται κατά βάση με δύο θέματα. Αφενός τον μηχανισμό επιλύσεως διαφορών και το άλλο στην τελευταία παράγραφο ή στις τελευταίες δύο παραγράφους τη ρυθμιστική συνοχή στην ίδια τη συζήτηση συχνά συζητείται με, με, με, με τρόπο που αμφισβητείται δηλαδή ο μηχανισμός επιλύσεως διαφορών. Γι' αυτό έχω περιλάβει στα έγγραφα, ελπίζοντας ότι μπορώ να συμβάλλω αντικειμενικά στη συζήτηση αυτή με την ερώτηση χρειαζόμαστε πράγματι τέτοιο μηχανισμό επιλύσεως διαφορών. Και στη δεύτερη ερώτηση, εφόσον απαντήσουμε καταφατικά δηλαδή, τι μορφή μπορεί να λάβει ένας τέτοιος μηχανισμός επιλύσεως διαφορών. Οι συζητήσεις που διεξάγουμε και έχουμε διεξαγάγει ήδη και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και με ανταλλαγή απόψεων στην τελευταία συνάντηση και εδώ ήταν πολύ σχηδής. Αφενός αναρωτηθήκαμε εάν αποδυναμώνει την δημοκρατία, αν μειώνεται το επίπεδο προστασίας, αν ο μηχανισμός αυτός οδηγεί και σε συμπεριφορές που κανονικά θα ήταν απαγορευμένες την χώρα του καθενός μας. Μπορεί ενδεχομένως να αντιθούν οι διαφορές από τα εθνικά δικαστήρια. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα θέματα εκεί. Κάτι που και νομικά δεν στέκει πάντα απόλυτα, όμως ακούεται μια κριτική και στην κοινή γνώμη, από πλευράς κοινή γνώμης δηλαδή, που κάπως πρέπει να απαντήσουμε σε αυτήν. δεν είναι δεδομένη εμπιστοσύνη στον μέχρι τώρα διατυπωθέντα μηχανισμό επιλύσεως διαφορών. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σε όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε να τα περιορίσουμε κάπως ώστε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όντως χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό επιλύσεως διαφορών. Στο ερώτημα αν τον χρειαζόμαστε ή όχι, για μένα το ερώτημα αυτό είναι λιγότερο σημαντικό διότι σε κράτη δικαίου πάντα μπορούν να λυθούν με δίκαιο τρόπο οι διαφορές. Δεν έχει νόημα δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους διεθνή συμφωνία μετά να αναφιούν προβλήματα και ο να μην γνωρίζει πώς επιλύονται τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να σκεφτούμε λογικά πρώτον ότι χρειαζόμαστε κάποιο μηχανισμό επιλύσεως διαφορών. Δεύτερο, να καθίσουμε να σκεφτούμε τι μορφή μπορεί να λάβει αυτός ο μηχανισμός επιλύσεως διαφορών. Έχω λοιπόν κάνει σχετικές προτάσεις στην πιο μακροχρόνια προοπτική θα πρέπει να πει κανείς ότι θα καταστεί αναγκαίο κάποιο δικαστήριο όπως συζητείτε τώρα άλλωστε στη Γερμανία τουλάχιστον. Ένα τέτοιο δικαστήριο λοιπόν θα ήταν λογικό. Βέβαια για να ιδρυθεί τέτοιο δικαστήριο δεν θα μπορέσει να θεσπιστεί αυτό. Δηλαδή δεν μπορέσει να πιάσει τόπο η ιδέα αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την συμφωνία TTIP. Γι' αυτό διατυπώνω στη γνωμοδότησή μου την πρόταση να προτρέψουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει με την σειρά της με ποιον τρόπο μπορεί να ιδρυθεί τέτοιο δικαστήριο το οποίο να εξοπλιστεί και με μηχανισμό προσφυγής σε δεύτερο βαθμό. Έτσι ώστε να αποκτήσουμε και τη γνώση για το πώς είναι δυνατό να δημιουργηθεί τέτοιο δικαστήριο μακροπρόθεσμα. Τώρα, για το τι μπορεί να ισχύσει ως μηχανισμός επιλύσεως διαφορών στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα, μέχρι ότου ενδεχομένως σε απότερο μέλλον δημιουργηθεί το δικαστήριο, το να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα, στο συμπέρασμα μάλλον ότι δεν θέλουμε να έχουμε κανένα μηχανισμό επιλύσεως ε, διαφορών, αυτό ε, νομίζω δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα, διότι ασφαλώς θα προκύψουν διαφορές. Και θα τεθεί το ερώτημα πώς θα επιληθούν διαφορέ διαφορές Ακούγεται και η ιδέα ότι θα μπορούσαν οι διαφορές αυτές να υποβληθούν σε διεθνή δικαστήρια. Εγώ προσπάθησα να το αξιολογήσω, να αξιολογήσω την ιδέα αυτή αντικειμενικά και νομικά. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν. Διότι ιδιώτες επενδυτές, ας πούμε, ιδιώτες δηλαδή γενικότερα, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε διεθνή δικαστήρια. Υπάρχουν τώρα ιδιαίτερες διεθνείς συμφωνίες που δεν είναι δυνατόν όμως να επεκταθεί η ισχύ τους ώστε να καλύψει και τα προβλεπόμενα από αυτή τη συμφωνία, διότι οι αρμοδιότητες αυτών των δικαστηρίων πάντοτε αναφέρονται σε τμήματα, όχι στο σύνολο των επενδύσεων, όχι στο σύνολο του ελεύθερου εμπορίου. Η ενιαία αγορά που έχουμε θεσπίσει εδώ είναι παρόμοια κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένα σημεία δηλαδή με μια ζώνη ελευθερών συναλλαγών. Και πάλι εκεί όμως τίθεται το ίδιο νομικό πρόβλημα της επιλύσεως των διαφορών. Θα μπορούσε επίσης ακούστηκε η γνώμη να γίνει διακρατικός η επίλυση της συμφωνίας δηλαδή η χώρα όπου έχει την έδρα του να σταθεί κατά της χώρας όπου έχει σημειωθεί η ε, ε, γενεσιουργός αιτία της διαφοράς. Αυτό όμως ασφαλώς θα οδηγήσει και σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Πώς θα προσφύγει ο ιδιώτης για προστασία του ατομικού του δικαιώματος σε διακρατικό επίπεδο. Άρα ούτε και αυτό αποτελεί λογική λύση. Συχνά ακούγεται η ιδέα επίσης ότι τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να αναλάβουν την επίλυση των διαφορών. Και εδώ όμως μπαίνουμε σε μια νομική συστημική προσέγγιση η οποία δεν είναι ασφαλής, δεν είναι όρθη. Διότι ξεκινούμε από μια διεθνή υπόθεση, καταλήγουμε μια διεθνή συμφωνία και καταλήγουμε σε μια εθνική δικαστική αρμοδιότητα. Τώρα, ατομικές υποθέσεις, οι ατομικές αποφάσεις για αυτές είναι αρμόδια τα εθνικά δικαστήρια. Για ένα είδος ωστόσο προσφυγής ενός ιδιώτη κατά ενός κράτους το να αχθούν ενώπιον του εθνικού, εθνικού δικαστηρίου μπορεί να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. Μπορεί να πει ο φυγόμενος ότι μου αρκεί το εθνικό δίκαιο, αλλά και πάλι τίθεται μια σχέση ανάμεσα στον ιδιώτη και στο διεθνές δίκαιο, όπου πάλι εκεί δεν είναι αντικειμενικά εξασφαλισμένη λύση. Γι' αυτό τίθεται το ερώτημα πάλι. Άλλωστε το εθνικό δίκαιο αποφασίζει σύμφωνα με το εθνικό τεθειμένο δίκαιο. Ενώ το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι αντικείμενο του εθνικού δικαίου. Έτσι λοιπόν με τη λύση αυτή των εθνικών δικαστηρίων πάλι την ανταποκρινόμεθα στις ανάγκες απονομής δικαιοσύνης. Μέχρι ότου υπάρξει ενδεχομένως στο μέλλον η θέσπιση ενός διεθνούς εμπορικού δικαστηρίου, κάτι το οποίο θα μπορούσε ως αρμοδιότητα να επεκταθεί και σε συστήματα αλλά θα χρειαστούμε ωστόσο ένα ενδιάμεσο μοντέλο. Άρα ένα μηχανισμό επιλύσεως διαφορών που να λαμβάνει υπόψη και τα υφιστάμενα προβλήματα και να μπορεί σε αυτά γι' αυτό εγώ προσπάθησα να σκιαγραφίσω μια τέτοια δομή που να λέει ότι δεν μένουμε στο επίπεδο ad hoc, στο εξειδικευμένο επίπεδο. Δηλαδή προσπαθούμε να επεκτείνουμε τα όσα ήδη έχουν προβληθεί στη Συμφωνία ΣΕΤΑ, να εξυγχρονιστούν όμως τα πράγματα αυτά και να εμπλουτιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί μηχανισμοί επιλύσεως διαφορών να περιοριστούν με τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να τα εξαλείψουμε. Βεβαίω, αν έχετε και εσείς κάποιες δικές σας ιδέες, πολύ ευχαριστώ, Αλλά μία δομή η οποία να εξασφαλίζει την αντιμετωπική αντιμετώπιση, να προσφέρει και μία δεξαμενή δικαστών, να έχει εξασφαλισμένη και μία, ένα τρόπο μάλλον αντιμετώπισης από πλευρά των δικαστών. Να μην υπάρχει ο φόβος ότι ενδέχεται να κατέλθουν κάποιες προδιαγραφές, να υπονομευθούν κάποιες προδιαγραφές. Να μην είναι δυνατόν αυτό δηλαδή. Μπορούν λοιπόν να βρεθούν τρόποι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση να δημιουργηθεί ο μηχανισμός επίλυσεως διαφορών, μπορούν να ευρεθούν οι τρόποι να αρθούν αυτές οι ανησυχίες μέχρι ότου να υπάρξει, μέχρι, μέχρι μάλιστα και να υπάρξει και βαθμός δικαιοδοσίας δεύτερος, δηλαδή προσφυγής στην, ε, κατά της απόφασης του πρώτου βαθμού. Ένα τελευταίο θέμα όσον αφορά την ρυθμιστική συνοχή. Επειδή και εδώ διεξάγεται συζήτηση ότι δηλαδή με τη ρυθμιστική συνοχή ενδεχομένως μπορεί να περιγραφεί η θέση, να καταστατηθεί η θέση του νομοθέτη. Θα πρόκειται για συνεργασία των συμβαλωμένων χωρών, αλλά σε ό,τι αφορά την υποβολή προτάσεων δεν θα μπορεί να αποκλείεται ποτέ ο νομοθέτης. Ούτε επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Και εδώ λοιπόν μπορούν να ευρεθούν κάποιες λύσεις και για να εξασφαλιστεί ότι τα προβλήματα να μην βασιστούν ούτε σε πολιτικό ούτε σε άλλο επίπεδο παρά μονάχα σε νομικό. Όπως είπα, ευχαριστώ να ακούσω άλλες ιδέες. Από τη δική μου σκοπιά πάντως πρέπει να αρθούμε νομίζω στο ύψος των περιστάσεων και νομίζω ότι η πρότασή μου μπορεί όντως να σας φανεί ε, ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ κύριε Κέσταρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας κύριε Φως. Το θετικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από την βούληση της εξασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εδώ λοιπόν πρέπει να είναι αυτό και το μέτρο της TTIP και το μηχανισμό επιλύσεων διαφορών. Δηλαδή, αν αυτό ο μηχανισμός διασφαλίζει την ευημερία της κοινωνίας και βελτιώνει τις προδιαγραφές προστασίας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Για τα διαιτητικά δικαστήρια έχω να πω κάτι τώρα. Βεβαίως τα εκτιμώ ιδιαίτερα κύριε αλλά σε ό,τι αφορά τους διαιτητές δικαστές, εκεί έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες τονίζουμε ιδίω την πτυχή ότι ιστορικά διαιτητικά δικαστήρια κρίθηκαν να κρίνουν ανάμεσα σε χώρες όπου από τη μια μεριά υπήρχαν αρχές κράτους δικαίου και από την άλλη μεριά όχι. Σε περιπτώσεις λοιπόν όπου δεν ίσχυαν αρχές κράτους δικαίου έπρεπε να υπάρχει κάποια εξασφάλιση για τις επιχειρήσεις που επένδυαν εκεί. Τώρα, στην συμφωνία TTIP έχουμε δύο οντότητες, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κράτη δικαίου. Άρα εκπίπτει εδώ ο λόγος για την θέσπιση διαιτητικών δικαστηρίων, τα οποία διαιτητικά δικαστήρια παραβιάζουν και μια βασική αρχή του κράτους δικαίου, ότι δηλαδή ο νόμος ισχύει Ισότιμα για όλους, Ισοδίκια για όλους. Έτσι εδώ ξεριζώνεται αυτή η βασική αρχή. Διότι έρχεται τώρα ιδιωτικό διαιτητικό δικαστήριο το οποίο δημιουργείται για χάρη των επιχειρήσεων. Για μένα αυτό αποτελεί μια κατάφορη παραβίαση των βασικών αρχών του κράτους δικαίου που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί ισοδίκια τα δικαιώματα όλων. Δεν χρειαζόμαστε ειδικά δικαστήρια για κάποιες ειδικέ ομάδες. Δεν χρειαζόμαστε για παράδειγμα ειδικά δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων ή των καταναλωτών ή ειδικά δικαστήρια για την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι τα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια δεν είναι κάτι που ενισχύουν, που ενισχύει τις αρχές του κράτους δικαίου. Δεύτερο, τα υφιστάμενα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια έχουν αδυναμίες. Είναι περιορισμένη η δημοσιότητα των συνεδριάσεών τους, δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεών τους και στη Συμφωνία ΣΕΤΑ εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Τέλος, σε αυτά τα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια στην ουσία οδηγούμεθα σε καταστρατήγηση των αρχών της δημοκρατίας όταν η έκδοση των αποφάσεων αφορά ιδιώτες. Γι' αυτό και συμφωνώ με τον πρώην συνταγματικό δικαστή Μπρος στη Γερμανία που θεωρεί ότι τα διαιτητικά δικαστήρια παραβιάζουν το γερμανικό σύνταγμα παραβιάζουν επίσης το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και μάλιστα λέει είναι και συστημική παραβίαση του ίδιου του διεθνούς δικαίου. Θεωρώ ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ διότι κινδυνεύουμε με τα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια να εκχωρήσουμε τμήμα της κρατικής κυριαρχίας σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα επιχείρημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και θέτω εν τέλει και το ερώτημα αν τα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια θα μπορούν να αντέξουν την κρίση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχω και μια τελική παρατήρηση για αυτήν την ρυθμιστική συνοχή. Εδώ καθίσταται προφανές ότι η αρχή αυτή της λήψης δημοκρατικών αποφάσεων από τα κοινοβούλια διότι νομοσχέδια θα συζητούνται σε ένα ξεχωριστό συμβούλιο και θα επηρεάζουν τη λειτουργία των ε, αυτό για μένα δεν συνάδει με τη λειτουργία των δημοκρατιών. Εδώ πάμε να δημιουργήσουμε μια δημοκρατία συμμορφούμενη με τις αγορές. Αυτό θεωρώ ότι είναι εσφαλμένη πορεία και για τις ΗΠΑ και για την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Η λοιπόν, Επιτροπή Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει τεράστια ευθύνη και θα πρέπει να εξετάσει πολύ διεξοδικά κάποια βασικά θέματα του TTIP, της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων. Και θα πρέπει για την εκπόνηση της έκθεσης μας, της γνωμοδότησης μας μάλλον, να αξιοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρογνωμοσία. Και χαίρομαι που ο κύριος Βάος εξετάζει και κάποιες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το ISDS, την επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή. Η ομάδα μου έχει τεράστιες επιφυλάξεις για την αναμορφωμένη πρόταση της επίλυσης διαφορών κράτους επενδυτού. Δεν νομίζω ότι έτσι ε, θα σεβαστούμε τις αρχές του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τι θα γίνει στο μέλλον. Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών που θα συμπεριληφθούν στο TTIP θα αποτελέσουν πρότυπο για πολλούς άλλους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Γι' αυτό και δεν θα, το πρέπει να, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα επιπόλαια ή ελαφρά την καρδία. Και μάλιστα όταν η ομάδα μου ανέλησε κάποιες υποθέσεις που θα στη, στον υπάρχοντα μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ISDS, διαπιστώσαμε ότι δεν ισχύει αυτό που ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι δηλαδή οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν εφαρμογή της νομοθεσίας. Πολλές επιθέσεις ε, ε, βάλουν κατά της νομοθεσίας. Στρέφονται κατά της ίδιας της νομοθεσίας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο επικριτική σε τέτοιες ε, δυνατότητες από ότι ο κύριος Φως. Γιατί ακριβώς αυτές οι δυνατότητες που διανοίγονται μας πείθουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά το εθνικό δίκαιο των συμβαλόμενων μωρών εφαρμόζεται και στο μέλλον δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ε, θα είναι κρίμα να μπορεί να αποσβητηθεί τέτοιο εθνικό δίκαιο από, επίλυση, από τέτοιο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα πολύ διεξοδικά για να βρούμε τη σωστή διαδικασία και το σωστό μηχανισμό. Ο κύριος Φως είπε κατά πόσο το σκόπιμο να θεσπιστεί ένα μόνιμο δικαστήριο. Ας το εξετάσουμε σοβαρά. Γιατί ο ισχύων μηχανισμός ISDS, ακόμη και με την μεταρρύθμιση που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι προσωρινή λύση μόνο, πώς θα μπορούμε στο μέλλον να, να τον αλλάξουμε. Γιατί πολλοί εμπειρογνώμονες διεθνούς δικαίου λένε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τα πιο ανεπτυγμένα νομικά συστήματα. Οπότε μπορούν ήδη να καλύψουν τέτοιες υποθέσεις και αγωγές επαιδητών, αλλαδαπών επενδυτών κατά του, του κράτους. Και ελάχιστα είναι τα κράτη που δεν έχουν αντίστοιχα ε, θέματα στα δικά τους νομικά συστήματα και ελπίζω να καλύψουν αυτά τα κενά. Αρχικά, μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κώστερ, μηχανισμοί τύπου ISDS χρησιμοποιήθηκαν για να προστατευτούν οι επενδύσεις αναπτυσσομένων χωρών, σε αναπτυσσόμενες χώρες μάλλον, σε χώρες δηλαδή που στερούνται ενός στιβαρού νομικού συστήματος. Αφορά δηλαδή θέμα ε, προστασία επενδύσεων ουσιαστικά αυτός ο μηχανισμός. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα προβλήματα που ανακύψουν από μια κανονιστική ρυθμιστική συνεργασία. Είχαμε σχετικά πρόσφατα μια ακρόαση στην οποία γινόταν η σύγκριση μεταξύ του Αμερικανικού και του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου. Και ίσως στο μέλλον να δημιουργηθούν προβλήματα στην κανονιστική συνεργασία μας. Συμφωνώ κύριε Φως με το ότι η έγκριση της εθνικής νομοθεσίας ε, θα πρέπει να γίνεται από νομοποιημένα νομοθετικά σώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Το θέμα είναι στο μέλλον θα ισχύσει αυτό. Γιατί φοβάμαι ότι το Σώμα Αριθμιστικής Συνεργασίας όπως έχει προγραμματιστεί ή όπως έχει σχεδιαστεί ίσως αναλάβει ε, σημαντικές εξουσίες και ίσως ε, προδικάζει κατά κάποιο τρόπο νομοθετικές προτάσεις και να υποκαθίσταται ουσιαστικά στην νομοθετική εξουσία. Να αντικαθιστά δηλαδή το Κογκρέσιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πού θα μπορούσε να οδηγήσει τέτοιου είδους κανονιστική συνεργασία. Πέραν του ISDS και της κανονιστικής συνεργασίας υπάρχει και μια τρίτη ιδέα στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κέστερ. Το θέμα της συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο, με το ενωσιακό δίκαιο και κατά πόσο τηρείται αυτό από τον ISDS. Λένε πολλοί νομομαθείς ότι η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου δείχνει ότι δεν είναι αυτονόητο ή αυταπόδεικτο ότι ο μηχανισμός ISDS ε, θα πληρεί τις προϋποθέσεις ε, του ενωσιακού δικαίου και του, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το ISD συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να διερευνήσουμε το θέμα πιο διεξοδικά. Γιατί η δική μας ε, Επιτροπή είναι αρμόδια με τη διαμόρφωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας Ευχαριστώ. Επιθυμείτε κύριε Φως να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ε, βέβαια δεν θα είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Εν τέλει έχω την αίσθηση ότι αυτό το θέμα πώς πρόχνουμε μπροστά μας. Θέλουμε να διαμορφώσουμε κάτι ή όχι. Το να λέμε μοναχά ότι είμαστε αντίθετοι και να περικόψουμε κάποια δικαιώματα του επενδυτού, αυτό είναι εύκολο, απλό. Αλλά ποια ακριβώς είναι η εναλλακτική επιλογή. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω. Για αυτόν που θα έλθει να επενδύσει χρήματα σε κάποια άλλη χώρα, τίθεται το ερώτημα πώς θα εξασφαλίσει τα δικαιώματά του με τον καλύτερο τρόπο. Καθαρά τώρα από άποψη συστημική, μια τέτοια σύμβαση που διαπραγματεύεται κανείς εδώ, συστημικά, δεν εντάσσεται στο εθνικό δίκαιο. Και επομένως δεν είναι δυνατόν ανεφετέρου να υπαχθεί στην δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηριών. Ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα. Στο διεθνές δίκαιο επίσης δεν είναι τόσο εύκολη η λύση. Γι' αυτό έχουμε μια δυτή κατάσταση εδώ, όπου δηλαδή το διεθνές δίκαιο έρχεται και τέμνεται με το ιδιωτικό δίκαιο. Γι' αυτό χρειάζεται κάποια διαμόρφωση ενός συστήματος από μέρους μας και μιας αρχής που λέει ότι μπορούν να δοθούν ορισμένα δικαιώματα στο άτομο για να λύσει κάποια προβλήματα αλλά είναι σαν να του λέει το εθνικό δίκαιο ότι τα προβλήματα που μπορεί να έχει δεν θέλω να τα κρίνω καν ή πάντω σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν σε δικαιώνει. Εάν εξετάσουμε τώρα την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Νότια Κορέα όπου αρχικά ήταν αρνητικό το ισοζύγιο των συναλλαγών αυτών με την Κορέα. Μετά από την θέσπιση και υπογραφή της συμφωνίας και τη θέση της σε ισχύ, το ισοζύγιο των συναλλαγών με την Κορέα είναι πλέον θετικό. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το θετικό πρόσημο πλέον του ισοζυγίου συναλλαγών ασφαλώς και έχει θετική επίδραση στην κοινωνική ευημερία της Ένωσης. Δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο, για παράδειγμα με την διατήρηση θέω απασχολήσω. Δεν ξέρω πώς, αλλά έχει κάποια θετική απήχηση στην ευημερία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αν θέλουμε τώρα να εξετάσουμε από συστημική νομική άποψη πώς θα αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις στο δικαιικό επίπεδο εάν δεν καταγραφεί ένα τέτοιο σύστημα στο, στη συμφωνία αυτή. Ο τεξανός δικαστής εκλέγεται για παράδειγμα και αυτός από τον ψηφοφόρο και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ανεξάρτητος. Όχι, δεν μπορούμε. Διότι δεν έχει νομικά την δυνατότητα να ελέγχει το διεθνές δίκαιο. Ανοίγουμε λοιπόν εδώ τον δρόμο σε διακρίσεις. Εάν απορρίψουμε την ιδέα λοιπόν αυτή του πιχαρισμού επιλύσεως διαφορών, πώς θα εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα του επενδυτού και αν ακόμα Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, εγώ θεωρώ, απέναντι στον ISDS δηλαδή, μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος να διαμορφωθεί δηλαδή το ενδεχόμενο αυτό διαιτητικό δικαστήριο έτσι ώστε είτε να ελαχιστοποιηθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα είτε και να αποκλειστούν εντελώς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να είμαστε ανοιχτοί, να καταδείξουμε και μια βούληση να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση κάποιου συστήματος διότι αλλιώς δεν βλέπω βούληση να προστατευτούν οι επενδυτές. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ρυθμιστική συνοχή, εμείς ως νομοθέτες δεν θεσπίζουμε βεβαίως και τις τελευταίες τεχνικές προδιαγραφές. Υπάρχουν οι οργανισμοί ΣΕΝ και ΣΕΝΕΛΕΚ, το Ινστιτούτο DIN στη Γερμανία των τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή της βιομηχανίας. Αυτά τα ρυθμίζουν αυτοί οι οργανισμοί. Δεν είναι λοιπόν θέματα τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς. Είναι λοιπόν το ερώτημα. Μπορούμε εμείς να πούμε ότι αντί του νομοθέτου κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, οργανισμοί βλέπε, ρυθμίζουν και θεσπίζουν επιμέρους προδιαγραφές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρείται κάτι από την αρμοδιότητα του νομοθέτου. Γι' αυτό και ξαναθέτω επιταπητώ το ερώτημα. Ποιες μπορούν να είναι οι εναλλακτικέ επιλογές. Κάτι που μπορεί να θεωρείται ως κακό ή έστω ανεπαρκές. Δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί με κάποιο τρόπο ώστε εν τέλει να εξυπηρετεί ο σκοπός της προσελκύσεως των επενδυτών. με ταυτόχρονη διατήρηση της αρχής της προστασίας των επενδυτών. Και αυτή η αρχή του, της ισότιμης εφαρμογής του δικαίου επί όλων, κύριε Κέστερ μα δεν επενδύουν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως αυτό που ενδιαφέρει είναι όλοι οι επενδυτές να την χάνουν ισοδίκης μεταχείρισης. Αυτά τα γράφουν και τα συντάγματά μας. Τα γράφει και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν τέλει και νομίζω ότι είναι λογικό αυτό που λέει η κυρία Χάουταλα, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη που να έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί στο μέλλον, ώστε να καλύψει και μελλοντικά πράγματα. Ίσως το διαιτητικό δικαστήριο να μην ήταν η απόλυτη λύση ως τώρα. Αν όμως το εξυγχρονίσουμε και το εξελίξουμε προς την κατεύθυνση ενός εμπορικού δικαστηρίου, τότε νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Και σε ό,τι αφορά αυτές τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που, τις οποίες αναφέρατε, υπάρχουν ήδη διμερείς συμφωνίες μεταξύ ε, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ενωμένων Πολιτειών. Δεν λέω βεβαίω ότι αυτές οι χώρες είναι λιγότερο ανεπτυγμένε, αλλά το νόημα της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών δεν είναι η επίλυση προβλημάτων. Το νόημα της ε, Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών είναι να διεξάγεται ελεύθερα το εμπόριο. Έτσι δεν είναι. Αλλά για την περίπτωση που αναφιούν προβλήματα να υπάρχει ένα μηχανισμό που να επιτρέπει την επίλυσή του. Θεωρώ λοιπόν ότι στην ουσία έχουμε στα χέρια μας και σε ό,τι αφορά την TTIP τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο να μπορεί να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί και στα σε ό,τι προκύψει στο μέλλον. Χωρίς να προβαίνουμε σε διακρίσεις βάρος κανενός. Διότι, διότι πρόκειται τελικά για την προστασία και την επίλυση του θέματος κάποιου ο οποίος επενδύει αλαχού. Λέω λοιπόν να προσεγγίσουμε το θέμα με κάποια θέληση διάπλασής του, διαμόρφωσής του. Να προχωρήσουμε με ένα μηχανισμό για να μπορούμε να διευκολύνουμε το ελεύθερο εμπόριο, το οποίο μας έχει ωφελήσει έως τώρα όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άντερσον, μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του. Ο εισηγητής επανειλημμένα αναρωτήθηκε ποια είναι η εναλλακτική ε, για την προστασία των ε, επενδύσεων και Είμαι περίεργος λοιπόν. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον εισηγητή ποια είναι η άποψή του σχετικά τα κατά όσον αφορά την ε, την ασφάλεια, την προστασία μέσω ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πριν απαντήσει ο εισηγητής, ε, θα πρέπει να σας πω ότι έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γκαρσία Βερθέρο, αναπληρωτής ε, διευθυντής της DG Trade. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε την δυνατότητα ε, να κάνω μερικά σχόλια ενώπιον της Επιτροπής σας ε, ως επικεφαλής διαπραγματευτής της εν λόγω συμφωνίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση για τη διατησία είναι μία από τις πιο κρίσιμες συζητήσεις ε, που πρέπει να κάνουμε στην TTIP και μάλιστα γίνονται σε μία κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια σχόλια λοιπόν από την οπτική γωνία της Κοπησιών έτσι ώστε να τις λάβετε υπόψη στην έκθεσή σας. Από την άποψη λοιπόν της Κομισιόν, ή ε, ε, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει διεθνής διαιτητική διεργασία στη συμφωνία, αλλά ε, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι μηχανισμοί διατησίας. Στις ε, πολυμερείς ε, συμφωνίες υπάρχουν αυτού του είδους οι προβλέψεις όσον αφορά την διατησία, ωστόσο δεν είναι κατάλληλες, είναι πλέον απαρχαιωμένες στον 21ο αιώνα. Επομένως θα πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί διατησίας που θα ανταποκρίνονται ε, στις ε, πραγματικές ε, υπερβολές και καταχρήσεις οι οποίες έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την διαιτησία σε περιπτώσεις επενδύσεων και διαφωνιών όσον αφορά τις επενδύσεις θα ε, ήθελα να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες ε, επαφές και συζητήσεις, αλλά παρόλα αυτά στο λίγο χρόνο που έχω θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια βασικά ε, στοιχεία. Πρώτον, η προστασία των επενδύσεων θα πρέπει να καθοριστεί με σαφή τρόπο έτσι ώστε να μην μπορεί να ε, ε, ε, παρουσιάζεται οποιοδήποτε κίνδυνο όσον αφορά τα ρυθμιστικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάναμε αυτό στην συμφωνία με τον Καναδά και προτείνουμε εδώ να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα στη συμφωνία με τις ΗΠΑ Δεύτερον, είμαι θα ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι διαιτητές υπό την ισχύουσα συμφωνία μονάχα οι διαιτητές οι οποίοι ε, ε, έχουν πραγματικά ε, προσόντα θα μπορούν, θα πρέπει να μπορούν να παρεμβάνονται στη διαδικασία διατησίας. Είναι κάτι το οποίο έχουμε υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι νομικοί έλεγχοι και οι απαραίτητοι μηχανισμοί έτσι ώστε σε περίπτωση που η διατησία δεν αποδίδει σε μικρό χρονικό διάστημα να υπάρχει έφεση σε άλλο επίπεδο. Ε, στη διαπραγμάτευση το συζητούμε αυτό γιατί αν ε, ε, μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία για το θέμα αυτό με τις ΗΠΑ τότε θα ανοίξουμε περιθώρια για μια γενικότερη, σφαιρικότερη μεταρρύθμιση του θέματος. Δεν έχω πολύ χρόνο έτσι ώστε να συζητήσω μαζί σας ακόμα περισσότερο, αλλά θα δραχθώ οποιασδήποτε ευκαιρία που μου παρουσιάσετε έτσι ώστε να συζητήσουμε το θέμα αυτό ξανά. Κύριε κυρία Φως, έρχομαι στην ερώτηση σας κυρία Άντερσον. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με τη δυνατότητα αντιμετώπιση από ασφαλιστικές εταιρείε. Βρίσκω ότι θα υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον από οικονομική σκοπιά, αλλά δεν αλλάζει και τίποτε ότι δεν είναι δυνατότητα προσφέρει το κράτο δικαίου. Ίσως τελικώς χορηγείται αποζημίωση στο οικονομικό επίπεδο, μπορεί να ικανοποιεί ίσως και τον επενδυτή, αλλά δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Ούτε ξέρω αν μπορούν να καλυφθούν όλες οι απαιτήσει του. Ομολογώ ότι δεν έχω εγκύψει βαθύτερα στο πρόβλημα, πρόκειται για, μόνο για μια πρώτη αυθόρμητη απάντηση. Μπορεί βέβαια ο επενδυτής, μπορεί ο επενδυτής να εξασφαλιστεί έτσι περαιτέρω με ε, σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά δεν έχει σχέση με την επίλυση του θέματος σε επίπεδο δικαίου. Είναι θέμα προσωπικής επιλογής, αλλά όπως το κατανοώ τουλάχιστον δεν είναι το ίδιο, δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Όπως λέω, μπορεί να είναι μια συμπληρωματική δυνατότητα να καλύψει τα νότα του και από άποψη οικονομική. Δεν μπορεί να αποτελέσει όμως πραγματική εναλλακτική επιλογή στην προστασία του επενδυτού καθ' αυτήν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος αυτού και προχωρούμε στο υπαριθμόν 8. Εξέταση σχεδίου εκθέσεως για το πρόγραμμα REFIT, βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας. Η κυρία Κάουφμαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα διεξαγάγαμε εκτεταμένη συζήτηση για το πρόγραμμα REFIT. Εκεί είχα αναπτύξει τις απόψεις μου, άρα δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, διότι άλλωστε έχει προχωρήσει και η ώρα. Επιθυμώ, μόνο να επενθυμίσω στις και στους συναδέλφους ότι σήμερα διαμορφώνεται διαφορετικά η κατάσταση από ότι την εποχή του Ιουνίου πέρσι όπου η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει το πρόγραμμα REFIT. Έχουμε τώρα νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος έχει ρητή αρμοδιότητα για θέματα βελτίωσης της ε, νομοθεσίας. Έχουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι στις 22 Τετάρτου θα υποβληθεί ευρύ πακέτο για την βελτίωση νομοθεσία από πλευρά τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι το REFIT θα συνεχίσει να είναι τμήμα του πακέτου αυτού που θα υποβληθεί στις 22 Τετάρτου και έρχομαι στο θέμα που είναι σημαντικό και για εσάς και για μένα Μέχρι τώρα δηλαδή παραπέμπω μόνο στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου 2014. Όμως ο καιρός περνά, στις 22 Τετάρτου θα λάβουμε το νέο πακέτο και για όλες και όλους εμάς, ιδίως όμως για εμένα ως εισηγήτρια, πρέπει να αναμένουμε ότι αυτά που αποτελούν τώρα αντικείμενο της ε, εκθέσεώς μου θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Αυτά θέλω να πω στις συναδέλφους μου και ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να τροποποιήσω το κείμενό μου εφόσον προκύψει νέα κατάσταση από την ε, επερχόμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε για σας και για μένα είναι σημαντικό τα πράγματα αυτά να είναι πλήρως ενημερωμένα. Και ενδεχομένως να αποδίδουν και κάποιες διαφορετικές νοηματικές αποχρώσεις. Θα ήθελα μόνο να πω, εάν εξετάσετε το κείμενο, είναι χωρισμένο σε 7 παραγράφους, περιλαμβάνω γενικά το ζήτημα της βελτίωσης της νομοθεσίας, της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το θέμα της μελέτης των επιπτώσεων, το ζήτημα των δοκιμασιών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της εκτονιστέρων αξιολογήσεως, το ζήτημα της λεγόμενης επιχρήσωσης ή της εφαρμογής των κανόνων από τις χώρες μέλη και τέλος το ζήτημα της απόσυρσης νομοθετικών προτάσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για όλα αυτά τα θέματα θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα. Από τη δική μου σκοπιά είναι για μένα σημαντικό ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσουμε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κομισιόν είπε ότι κατευθύνεται σε νέα διαθεσμική συμφωνία με Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών, κάτι το οποίο από καιρού ζητεί το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι επιθυμούμε να πορευθούμε μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα σε αυτή την πορεία και θεωρώ ακόμη ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν πρόκειται τόσο για τον αριθμό των νομοθετημάτων, για την ποσότητα δηλαδή, αλλά για την βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας. Όταν 28 χώρες μέλη θεσπίζουν από κοινού μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, αυτό, η προσπάθεια αυτή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της γραφειοκρατίας αφού θα αντικαταστήσει 28 ξεχωριστές κρατικές ρυθμίσεις. Για τα τεστ των ΜΜΕ χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει αυτές τις ε, δοκιμασίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως γνωστόν είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας και είναι σωστό να μειωθεί το ε, γραφειοκρατικό βάρος που αντιμετωπίζουν το ίδιο. Σημαντικό είναι και είναι προς το συμφέρον όλων να φροντίσουμε ώστε η μείωση του γραφειοκρατικού βάρους να μην σημάνει και μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να είναι εξασφαλισμένα. Είναι σωστό που η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της περί Refit αναφέρεται σε αυτό και λέει ότι σαφώς αυτό δεν αποτελεί στόχο της να πω τώρα κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μένα, στην τελευταία παράγραφο, δηλαδή απόσυρση νομοθετικών προτάσεων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ εμπλέκονται και τα δικαιώματα του Ευρωκοινοβουλίου. Η πρώτη, για πρώτη φορά μάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και όπως γνωρίζετε έχει κάνει πολλές προτάσεις αποσύρσεως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε όμως ότι δεν συμφωνεί με όλα. Κάναμε μια ψηφοφορία τον Γενάρη όπου είπαμε συγκεκριμένα ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιθυμούμε να αποσυρθούν ορισμένα νομοθετήματα. Εδώ οδηγούμεθα σε μια σύγκρουση σε επιμέρους θέματα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εγώ επεσήμανα στην έκθεσή μου ένα πρόβλημα που μου φαίνεται σημαντικό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αποσύρει νομοθετικές προτάσεις με την παρατήρηση ότι δεν προβλέπεται συνένεση στο Συμβούλιο Υπουργών. Εμείς όμως ως συνομοθέτης έχουμε ήδη τοποθετηθεί και θεωρώ ότι εάν το καλοψάξουμε βλέπουμε να υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στα δύο σκέλη του νομοθετικού. Δεν λαμβάνονται δηλαδή επαρκώς υπόψη τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Αυτό μου φαίνεται εμένα κέρια σημασίας σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας και αυτά πρέπει να τα διαπραγματευτούμε στο μέλλον με Συμβούλιο και Κόμισιον. Διαπιστώνω επίσης ότι στο γερμανικό κείμενο στις παραγράφους 22 και 28 έχουν παρισφρήσει κάποια ίσον ασφάλματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μου είπαν ότι το αργότερο αύριο μεθαύριο θα έχει διορθωθεί το κείμενο στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ λοιπόν που με ακούσατε. Αναμένω με μεγάλη χαρά τη συνεργασία μαζί σας. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι η 34 δηλαδή μία εβδομάδα μετά από την υποβολή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Εκεί θα δούμε τότε ποια ίσως ακόμα πράγματα θα πρέπει να περιλάβουμε στο κείμενό μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου σε μεγάλο βαθμό είναι ικανοποιημένη με το σχέδιο έκθεση Κυρία Κάουφμαν και είναι σημαντικό αυτό που είπε ότι ούκαν το πολλό το F, το τα αφορά την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Και έχει νόημα εκεί που ένα κοινοτικό νομοθετικό μέτρο μπορεί να αντικαταστήσει 28 εθνικά. Συμφωνώ με την προσέγγιση της συγγήτριας ότι η αρχή της πολιτικής ασυνέχειας που χρησιμοποιεί αρκετά συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποσύρει προτάσεις της δεν ενισχύει τη συνεργασία ή την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε στις αρμο... Θα πρέπει να το συζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αρμόδιες επιτροπέ περιλαμβάνουν τέτοιε αποφάσεις. Επίσης, οι μελέτες επιπτώσεων δεν υποκαθιστούν τι πολιτικέ ε, αξιολογήσει. Είναι σημαντικές ε, οι μελέτες επιπτώσεων, αλλά δεν είναι θέσφατο. Ε, οι πολιτικοί θα λάβουν την τελική απόφαση. Είναι θέμα πολιτικής αξιολόγησης, τελική ανάλυση. Συμφωνούμε με την έμφαση που δίνει η κυρία Κάουφμαν στον διάλογο μεταξύ των δύο βραχιώνων της νομοθετικής αρχής και μεταξύ αυτών και των πολιτών. Αύριο θα έχουμε μια εκτακτή δημόσια ακρόαση για κάτι που κατά τη γνώμη είναι το πιο αναποτελεσματικό νομοθετικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η οδηγία για τη θερινή ώρα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκούτελαντ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Κάουφμαν. για το σχέδιο που μας υπέβαλε. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό που επισήμανε η εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή, Επιστροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι πρέπει να αποσύρει κάποιες νομοθετικές προτάσεις, είτε γιατί είναι περίπλοκη η νομοθετική διαδικασία, είτε γιατί θα ήταν ευκολότερο να καταργήσουμε ή να μην διωγγώνουμε το νομοθετικό μας έργο. Δεν νομίζω ότι εφταθούν αυτά τα δύο επιχείρηματα. Το πρώτο επιχείρημα της περίπλοκης διαδικασίας ε, δεν ισχύει, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να αντιμετωπίζει και μελλοντικά προβλήματα. Τέτοια θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το δεύτερο επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι καλό θα ήταν να αποσύρει μερικές νομοθετικές προτάσεις για να μην ε, πολλαπλασιάζει τις νομοθετικές ρυθμίσεις και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, γιατί αυτά τα επιχειρήματα ακούμε. Εγώ πιστεύω και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είμαι μέλος και στην δική μας την Νομική Επιτροπή ότι ακριβώ η φιλοπεριβαλλοντική νομοθεσία, η νομοθεσία για το περιβάλλον έχει πληγεί από αυτή την προσπάθεια πλούστευσης ή μείωσης της νομοθετικής πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα δίστα πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση των επιχειρήσεων αν συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οπότε ούτε την πρόοδο νομοθετική πρωτοβουλία πρωτοβουλιας ευρωπαικης επιτροπης και μαλιστα θα Ένωσης εξυπηρετούμε, για συγκεκριμένε προδιαγραφέ. οποτε ουτε την προοδο διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις με την απόσυρση νομοθετικών προτάσεων. Και Χαίρομαι που το ζήτημα αυτό επισημάνθηκε και εδώ. Ευχαριστώ κύριε Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εγώ επιθυμώ πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για την έκθεσή της, για το σχέδιο εκθέσεως. Διαπιστώνω ότι έχει συμπεριλάβει πολλά πράγματα στην έκθεσή της, με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Χαίρομαι που προχωρεί πρώτα σε μια καταγραφή για το θέμα Refit δεν ε, περιλαμβάνει ξανά όλα τα σχέδια προτάσεων, άλλωστε δεν θα ήταν κάτι τέτοιο στόχος της εκθεσής της. Υπάρχουν και πολλά επιμέρους θέματα, κυρία Κάφμαν, όπου συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ορισμένα για παράδειγμα, άλλες συνάδελφοι είπαν ήδη ότι όντω πρέπει να ρίξουμε περισσότερο βάρος στην ποιότητα και λιγότερο στην ποσότητα των νομοθετικών προτάσεων. Συμφωνώ απολύτως, άλλωστε, αλλά έχω δουλέψει και πολλά χρόνια γι' αυτό. Δηλαδή, να βελτιστοποιήσουμε και τις δικές μας μελέτες επιπτώσεων του Κοινοβουλίου, να απευθύνουμε έκκληση και στις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό και αυτά που λέτε για το impact assessment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης με βρίσκουν σύμφωνοι, δείχνουν άλλωστε και πόσο σημαντικό είναι ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τα, ε, μιλώ για τα τεστ των ΜΜΕ και αυτά που είπατε για τις χώρες μέλη, δηλαδή να ξεφύγουν πλέον από αυτή την επιχρήσωση, από αυτό το gold plating και να μην φορτώνουν τις οδηγίες με παραπάνω πράγματα. Αυτά όλα τα, σε αυτά όλα συμφωνώ. Υπάρχουν δύο θέματα όπου ε, διαφωνώ στο κάτω της γραφής, χρειάζεται και η διαφωνία για να μην βαριόμαστε, ιδίως στην παράγραφό σας υπαριθμών 30, μου φαίνεται ότι το πρόγραμμα της ε, Κομισιόν είναι φιλόδοξο και κάνει πλέον τα λόγια της έργα, βγήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως και είπε ότι θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή θέλει να περιοριστεί στα ουσιώδη να ξεφύγει από τις υπερβολικές, υπερβολικά λεπτομερείς ρυθμίσεις. Εμένα μου φαίνεται ως αρχή σωστό αυτό και δεν το επικρίνω. Αντίθετα χαίρο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στα σοβαρά με την προσπάθεια αυτή. Η πρότασή σας να ενισχυθούν τα προνόμια των κοινωνικών εταίρων, αυτό, σε αυτό απέναντι εγώ στέκομαι κριτικά. Αλλά κατά τα άλλα επαναλαμβάνω ότι στην έκθεση σας περιλαμβάνεται πολλά και σημαντικά θέματα Κάποια που ίσως θα θέλουμε να συμπληρώσουμε ως πολιτική ομάδα θα τα περιλάβουμε σε τροπολογίες, ιδίως σχετικά με το ποια συγκεκριμένα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα η βελτιωμένη νομοθεσία. Έχουν κάνει οι συναδελφοί μου προεργασία. Εγώ συμφωνώ με τη ρύθμιση one in, one out και στις οδηγίες να μπαίνουν και καταληκτικές ρήτρες, sunset clauses. Αυτό οφείλουμε να το ζητούμε ως νομοθέτες και να ελέγχουμε και ε, με μέτρο αυτό τις νομοθετικές μας προτάσεις. Το θέμα επίσης που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον και που θα πρέπει ίσως να συζητηθεί εντατικά και με τις άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές, αυτό το ζήτημα της ασυνέχειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. που εδώ σε εμά δεν ισχύει και οι συνάδελφοί μου τη Γερμανική Bundestag έχουν ε, κάνει καλές εμπειρίες με αυτή τη δική μα στάση. Θα μπορούσε να ισχύσει αυτή η ασυνέχεια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ωστόσο. Γιατί έχουμε για παράδειγμα 60% νέους ευρωβουλευτές στο παρόν Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί αυτοί να δεσμεύονται από τα όσα έχουν προτείνει και αποφασίσει οι προηγούμενοι. Χαίρομαι λοιπόν που θέτετε το θέμα και στην έκθεση σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Α, η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. κύριε Πρόεδρε. Δύο στοιχεία συμπληρωματικά. Σημειώνω αυτή την 22 η Απριλίου που ε, ανέφερε η συγκητρια και που ενδεχομένως εκεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τώρα για το gold plating επιθυμώ να το τονίσω. Βεβαίως είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η συγγήτρια. Επιθυμώ ωστόσο να τονίσω ότι σε πολλούς τομείς της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής νομοθεσίας ομιλούμε για ελάχιστα στάνταρτ Ελάχιστε προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το gold plating, δηλαδή ο υπερθεματισμός. Μπορούν οι χώρες μέλη να θέλουν να βελτιώσουν τις αρχές αυτές. Ελάχιστε προδιαγραφές σημαίνουν ακριβώς ένα κατόφλι. Αν θέλουν τώρα να προχωρήσουν στο εθνικό επίπεδο, ε, δεν μπορεί να πει κανεί στις χώρε αυτέ, τίποτε άλλο παρά συγχαρητήρια. Άρα εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε τι σημαίνει η εφαρμογή ένα προς ένα, λέξη προς λέξη δηλαδή, της οδηγίας. Εάν την υπερβούν δεν είναι κακό απαραίτητα, αντίθετα αποτελεί μια περαιτέρω εξέλιξη, ειδικά ε, μιλώ για τις κοινωνικές και για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Το δεύτερο που θέλω να θέσω αναφέρεται σε μια από τις ε, περιπτώσεις εκείνες τις συμβάσεις των κοινωνικών εταίρων. Ε, βλέπετε συλλογικέ συμβάσεις όπου αυτό που προβλέπετε είναι εκείνοι οι οποίοι σε ορισμένου τομεί γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για την ε, πραγματική ζωή, για την πράξη, δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτοί να μπορούν, να πρέπει μάλιστα, να συμφωνούν να υπάρξει και μια ε, συνολική ευρωπαϊκή συλλογική σύμβαση ανατομέα. Αυτό πραγματικά ξεπηδάει μέσα από τη ζωή. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει περισσότερο σαν αυτή η δυνατότητα των εταίρων να πηγαίνει να περιοριστεί. Βέβαια θα χρειαζόταν αναθεώρηση της ε, συνθήκης της λειτουργίας της Ένωσης και αυτό δεν το βρίσκω ρεαλιστικό. Αυτό που διαβλέπω όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί βήμα-βήμα σε μια περικοπή των δικαιωμάτων των ε, κοινωνικών εταίρων να συμφωνούν. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Βλέπουμε επίσης όλο και περισσότερο δημόσιες διαβουλεύσεις επιγραμμικά, online δηλαδή, στο διαδίκτυο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Προσοχή λοιπόν. Οι δυνατότητε αυτές που υπάρχουν υπέρ των κοινωνικών εταίρων υπάρχει κίνδυνος με, με αυτή τη σαλαμοποίηση τελικά να αποδυναμωθούν. Ίσως να μην έχει έρθει βέβαια ακόμα το σωστό χρονικό σημείο για να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά σε αυτά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, οδηγούν μοναχά σε βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας, καμιά φορά οδηγούν και στο αντίθετο. κυρία Χάνιμπολ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί, αλλά στο τελευταίο κομμάτι ε, της ε, έκθεσης βλέπω όλα αυτά τα θέματα του τελευταίου τμήματος πολύ ανησυχητικά και πρώτη φορά συμβαίνουν μάλιστα. Νομίζω όσον αφορά την απόσυρση νομοθετημάτων η αρχή της πολιτικής λύσης της συνεχείας ε, το αναφέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τι θα, τι γίνει με το Κοινοβούλιο αυτή η απόρριψη κρεμουσών προτάσεων έχει ε, γίνει αποδεκτή από το Κοινοβούλιο ας πούμε το θέμα των ε, αδειών για τις μητέρες είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές αλλά δεν θα πρέπει να γίνει μια κανονική συζήτηση γι' αυτό

Ε, και οι απόψεις του Κοινοβουλίου θα πρέπει πραγματικά να λαμβάνονται υπόψη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Τώρα, εάν έχει συζητηθεί και έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, ε, εντάξει, ε, και ενδεχομένως συμβαίνει ή μπορεί να συμβεί αυτό που συμβαίνει και σε μερικές χώρες μέλη, δηλαδή ότι προηγούμενες αποφάσεις κοινοβουλίων μπορεί να δεσμεύουν επόμενα κοινοβούλια, εντάξει, αλλά νομίζω ότι εδώ τα πράγματα δεν αναφέρονται καλά και νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το ε, θέμα αυτό ε, και το σημείο της ε, έκθεσης γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ακρογωνίως λήθος στην πρόταση της Κομισιόν. Όταν το Κοινοβούλιο έχει περάσει αυτές τις εκκρεμούσες προτάσεις και οι οποίες παραμένουν εκκρεμείς λόγω λιγορίας της Κομισιόν, τότε δεν είναι δυνατόν να αποσύρονται οι προτάσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο λόγο στην Κομισιόνα, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σύμφωνα ε, με τη διατύπωση. Η Κομισιόνα έχει το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε πρόταση. Έτσι αναφέρεται ε, στις ε, συνθήκες και αυτή είναι η νομική κατάσταση. Ίσως δεν μας αρέσει, ίσως είναι ατυχής, αλλά παρόλα αυτά έτσι είναι. Η Κομισιόν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα κάνω πολύ, μερικά πολύ σύντομα σχόλια, 4-5 το πολύ. Ε, πρώτον, ε, ξεφύγαμε λίγο χρονολογικά, περιμένουμε η δέσμη να έρθει στις 28 Απριλίου και όχι στις 22. 28 Απριλίου. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα του Refit, ε, θα ε, ε, επαναλαμβάνω εντόνως ότι μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την προστασία των πολιτών και όχι να την μειώσουμε και δεν θέλουμε καθόλου να μειώσουμε τα πρότυπα. Όσον αφορά τώρα ε, τα υπόλοιπα θέματα, δεν μπορώ να σχολιάσω ήδη ένα πακέτο για καλύτερη νομοθέτηση το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει αλλά παρόλα αυτά λαμβάνονται υπόψη ε, πληθώρα μελετών ε, στην Κομισιόν και από κοινού η Κομισιόν με το Κοινοβούλιο θα ε, συζητήσει τα θέματα αυτά προς κάποιο συντονισμός. Επίσης ε, η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Βεβαίως εμείς συμμεριζόμαστε τα αναφερόμενα στο ε, σχέδιο ψηφίσματος. Ε, θέλουμε συζήτηση και με τα Κοινοβούλια. Αυτό που λέμε απλώς είναι ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν πολύ διαφορετικά συστήματα και σε μερικές περιπτώσεις τα Κοινοβούλια δεν αναμειγνύονται σε διαδικασίες τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Εθνική Διοίκηση διοίκηση. Βεβαίως θέλουμε να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο στενά με τα κράτη-μέλη για την ε, ε, εφαρμογή, την υλοποίηση των, ε, του νομοθετικού πλαισίου γιατί δύο, μερικές φορές ο τρόπος με τον οποίο σε ορισμένα κράτη-μέλη εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία προκαλεί αγγυλώσεις, τις οποίες βεβαίως δεν επιθυμούμε. Ε, και θέλουμε με κάποιο τρόπο να είναι πιο ομοιογενής η αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη της ενωσιακής νομοθεσία και να είναι πιο ομοιογενής η ε, ε, εφαρμογή. Επίσης, δύο θέματα να πω. Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι απέναντι στο Κοινοβούλιο να επεξηγούμε οποιαδήποτε απόσυρση αποφασίσουμε και δεύτερον ε, να περιμένουμε απάντηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων σε γενικές γραμμές είπε ότι ε, καλωσορίζει την πρόταση της Κομισιόν και δεν θα κάνει επιμέρους σχόλια. Καταλαβαίνουμε ότι το Κοινοβούλιο, είχαμε καταλάβει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει ε, ε, έκθεση ή ε, ψήφισμα για τα θέματα αυτά και γι' αυτό προχωρήσαμε στην απόσυρση και στην αναγγελία της απόσυρσης προτάσεων. Επίσης, ε, έχει ήδη ξεκινήσει, όπως είχε συμφωνηθεί η Κομισιόν, ε, όπως έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια της Επιτροπής Γιούγκερ, τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ε, έτσι ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να προχωρήσει αυτή η εργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο τελευταίος μας ομιλητής από το κατάλογο. Δεν ξέρω αν η κυρία Κάουφμαν θέλει να επανέλθει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, πολύ σύντομα επιθυμώ να επανέλθω. Πρώτα τα βεβαίως όλες τις συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και μου έθεσαν υπόψη τα σχόλιά τους. Θα επανέλθω στο θέμα της ασυνέχειας και της απόσυρσης νομοθετικών προτάσεων. Η κυρία Νίμπλερ αναφέρθηκε στην παράγραφο μου παριθμών 30. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε επ' αυτού. Πράγματι, δεν έχουμε εκδώσει ψήφισμα για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε όμως ψηφοφορία στην Ολομέλεια, όπου έχουμε τοποθετηθεί για επιμέρους νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπου είπαμε ότι αυτές δεν επιθυμούμε να αποσυρθούν τις περιλαμβάνουμε, τις περιλαμβάνω δηλαδή εγώ στην παράγραφό μου αριθμός 30. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποσύρει νομοθετικές προτάσεις της, ακόμα και αν έχουν ήδη γίνει αντικείμενο επεξεργασίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ταυτόχρονα έχουμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2010 που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει διόντως υπόψη την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίω, πρόκειται και μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο συνεργαζόμενα θεσμικά όργανα. Περί αυτού πρόκειται άλλωστε που επιθυμώ να τονίσω, ότι δηλαδή πράγματι οφείλει να ληφθεί υπόψη η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, αφού έχει τοποθετηθεί μάλιστα η Ολομέλεια. Και το ερώτημα είναι πώς, πού πάμε παρακάτω. Η επισήμανση τώρα της Κομισιόν, του εκπροσώπου της Κομισιόν, ότι η δέσμη θα υποβληθεί στις 28 Τετάρτη και όχι 22 όπως νόμιζα, για μένα θέτει ένα ερώτημα βεβαίως για την κατάθεση τροπολογιών, διότι αυτό θα σημαίνει ότι και εγώ και οι συνάδελφοί μου δεν θα έχουμε παραπάνω από δύο μέρες για να υποβάλουμε τροπολογίες. Τότε λοιπόν η υποθεσμία μας είναι πολύ σύντομη, υπερβολικά σύντομη. Θα έλεγα να παραταθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά από την κατάθεση του, της τη της Κομισιόν, δηλαδή της ανακοινώσεως της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και να ζητήσω από τον κύριο Καβαδά τον Αντιπρόεδρο να αναλάβει την Προεδρία για το επόμενο σημείο γιατί εγώ είμαι ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Οπότε θα ε, ανακουφίσουμε τη συνείδηση, θα απαλλάξουμε από τον πρόεδρο από την Προεδρία για να μπορεί να αφοσιωθεί στο έργο του που είναι να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Και τώρα θα σας μιλήσω τσεχικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω συντομία το σχέδιο την πρόταση ψηφίσματο σχετικά με την επιδίωξη ενωμένη συνένεση όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία στην εσωτερική αγορά. Σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο δράση περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Πιστεύω ακράδαντα ότι ε, θα έχουμε αρκετό χρόνο για την μελλοντική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση αυτών των δικαιωμάτων ε, εγώ εδώ ασχολούμαι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και θέλει να αντιδράσει στις σημαντικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στον τομέα αυτό. Μάλιστα, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση, δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους ιδιώτες ή να ποινικοποιήσουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές, απλώς ε, να αποτρέψουμε τον αθέμητο πλουτισμό που οφείλεται σε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Γίνεται μία ανάλυση της κατάστασης ε, και με διαβουλεύσεις ε, θέλουμε να, να δημιουργήσουμε πιο εμπεριστατωμένη γνώμη για την κατάσταση που επικρατεί και το πλαίσιο που ισχύει για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της, των εξτρατιών ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Βέβαια αυτά, αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι στοχευμένες και πολύπλευρες ώστε να εξοικειωθεί καλύτερα ο κόσμος με τα θέματα αυτά. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συμβάλλουν τα μάλα στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία νέων, θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό και θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη μου, έχει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις συγκεκριμένες μορφές στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, ε, κάτω τη συζήτηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις επιγραμμικές συναλλαγές, τις δυνατότητες που μας δίνει το διαδίκτυο. Γιατί πολλές παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας γίνονται μέσω διαδικτύου. Θα ήθελα με το ψήφισμα να διαβεβαιώσω και τους σκιώδης ηγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους ότι θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω ένα ευρύ φάσμα απόψε και περιμένω τα σχόλιά σας. Επειδή έχουμε ακόμη τρία σημεία στην ημερήσια διάταξη, θέλω να επιταχύνουμε λίγο τη συζήτηση. Κυρία Λεγκρίπ, είστε η πρώτη που έχετε το λόγο. Παρακαλώ, χρόνου φίδου. Και μετά ο κύριος Κόστινας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο Σφόμποντα για το ψήφισμά του. Πραγματικά είναι επιτακτική και κατεπίγουσα ανάγκη η χάραξη πολιτικής ε, για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη ότι η πρόθεση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σημαντική επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη. Γι' αυτό και θα πρέπει να βρούμε σαφείς και αποτελεσματικές λύσεις. Αυτό χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους δημιουργούς και τους εφευρέτες μας. Χαίρομαι που στην έκθεσή σας αναφέρετε συγκεκριμένες προτεραιότητες, τις οποίες εστερνίζομαι. Μιλάτε για ανάμειξη όλων των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για να αποφευθεί παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης θέλετε να καταπολεμήσουμε την παραποίηση και την πειρατεία αξιέπαινα και μιλάτε για το καθήκον της δέουσας επιμέλειας που θα πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να παταχθεί η παραποίηση. Μιλάτε για τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωση των καταναλωτών για να αφυπνιστεί το κοινό και να δει πόσο η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι επιζήμια και επίση αφιερώνεται και ιδιαίτερο κεφάλαιο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, επηρεάζονται από το θέμα αυτό και δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να αντιμετωπίσουν πιθανέ παραβιάσεις των δικών του δικαιωμάτων πνευματικής Αν Άμα επιτρέπετε μια πολύ μικρή επιφύλαξη, αλλά πραγματικά ίσορο σημασία. Στις παραγράφους 8 και 9 μιλάτε για μια σχέση κατά τη γνώμη αιτίου αιτιατού, κάπως όμως ε, ε, σε ό,τι αφορά την έλλειψη ανταγωνιστικής σχέσης ε, μεταξύ νόμων και παράνομων προϊόντων και μερικές φορές την στροφή του καταναλωτού προς παράνομα προϊόντα. Ίσως τη διατύπωση θα πρέπει να προσέξουμε εκεί για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, γιατί πιστεύω ότι και πολλές χώρες αλλά και πολλοί τομείς επικεντρώνονται στην ε, προσφορά νόμιμων προϊόντων και περιεχομένου. Γι' αυτό αυτή η σχέση αιτίου και αιτιατού που υποδεικνύεται ε, ίσως ε, δεν ευσταθεί. Κύριε Κώστα, παρακαλώ, εν συντομία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σόβοντα για την έκθεσή σας. να λάβουμε υπόψη τα εξή με το EU Action Plan. Πρώτον, μια πραγματική ισορροπία ανάμεσα στους πελάτες και στους δικαιούχους. Κάπως πρέπει να βελτιωθεί η ισορροπία στην πρόταση, ιδίως για να ενισχυθεί η προστασία των ιδιωτών πελατών. Θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο επίσης την αρχή follow the money. Έχω κάποια ερωτηματικά όσον αφορά την αρχή αυτή και μήπως αυτή οδηγεί ώστε η προστασία των συμφερόντων των ιδιωτών χρηστών πάνε να μειωθούν. Με αυτή την αρχή του ακολουθώ το χρήμα εισάγονται κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν την ελευθερία χρήση του διαδικτύου από την πλευρά των χρηστών δηλαδή. Να προσέξουμε επίσης όταν μιλούμε για ποινικέ διώξεις όπως την έκθεσή σας κύριε Σφόβοντα μην οδηγήσουμε σε μια μην προωθήσουμε δηλαδή την ε, εγκληματικοποίηση των χρηστών, να το πω έτσι. Στο σχέδιο δράσης λαμβάνονται υπόψη ιδίω τα δικαιώματα των δημιουργών. Σημαντικό αυτό, γιατί γίνονται περικοπές τώρα και στον τομέα του πολιτισμού. Το Action Plan πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα των δημιουργών στον χώρο της τέχνης. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι χρειαζόμαστε αξιόπιστες, αξιόπιστους ελέγχους και αξιόπιστα δεδομένα για τις βλάβες που υφίστανται οι δικαιούχοι. Οι μελέτες που έχουμε δεν είναι αξιόπιστες έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια πραγματικά στέρεη, αξιόπιστη αξιολόγηση των επιπτώσεων, των δυσμενών επιπτώσεων της παραβιάσεως του δικαίου αυτού. Ε, κύριε Αντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη λαμβάνοντας υπόψη την ώρα. Θα ήθελα βεβαίως να συγχαρώ τον εισηγητή και πρόεδρό μας. Θα ήθελα μονάχα να εκφράσω μια μικρή δυσφορία. Δεν θέλω να ποινικοποιούνται αυτοί που δεν σέβονται απολύτως και πάντα ε, τα διευνητικά δικαιώματα, αλλά βρίσκω ότι υπάρχει ε, υπάρχει μία έτσι ε, πολύ μεγάλη Η υπερβολική επίοικια για αυτού που παραβιάζουν συστηματικά ε, την ε, πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη δημιουργία. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να θεσμοθετήσουν αυτή την παραβίαση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Άντερσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του. Δεν θα την είχα ακριβώ γράψει έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω ότι είναι μια καλή προσπάθεια για ισορροπημένη έκθεση. Θα υποβάλουμε άλλωστε τροπολογίες έτσι ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εργασία αυτή, ενδεχομένως ε, και ευελπιστώ μέσω συμβιβαστικών λύσεων. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είμαι πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ να μιλήσω στα αγγλικά. Επομένως θα υποβάλω τις τροπολογίες μου και ευελπιστώ ότι θα τις δεχτείτε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέμβαση. <laughs> Γιατί λαμβάνοντα υπόψη το προκεχωρημένο τη ώρα, το καλύτερο. Ναι, χρειαζόμαστε και λίγο χιούμορ. Η Κομισιόν θέλει οπωσδήποτε να μας ε, ε, πει δύο λόγια. Ε, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βερζερού, σας παρακολουθώ στενά. Δύο λόγια μονάχα έτσι ώστε να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Όσον αφορά το follow the money, καθόλου δεν είναι να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα στραφεί εναντίον ατόμων. Θέλουμε να υπάρχει ιδέουσα επιμέλεια έτσι ώστε να αποτραπούν κάποιες ε, παραβιάσεις και ε, ε, επομένως να ε, δίνεται η άδεια για ε, πρόσβαση σε προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας ε, αλλά με προστασία απέναντι σε παραποιημένα προϊόντα, απέναντι σε προϊόντα τα οποία έχουν παραβιάσει τη διανοητική ιδιοκτησία κτλ. Δεν υπάρχει καθόλου καμία πρόθεση να περιορίσουμε τον τελικό καταναλωτή. Πέραν αυτού, πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος συγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πήρα ένα μάθημα για το πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τη συζήτηση. Μερικές μέσα απαντήσεις τώρα. Ευχαριστώ για τις τροπολογίες σας, τις οποίες θα συμπεριλάβω στην έκθεση. Ό,τι αφορά την ποινικοποίηση που είπατε κάποιων δραστών παραβατών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το, πνευματικό, το ποινικό συγγνώμη δίκαιο προβλέπει δόλο κατά τη διάπρεξη ενός εγκλήματος και αυτό το λαμβάνω υπόψη και εγώ. Πουθενά δεν λέω ότι είναι θεμητή η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Αν έδωσα αυτή την εντύπωση ήταν παρεξήγηση πραγματικά και με τι τροπολογίε σα θα τη διορθώσω. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να παραβιάσουμε ούτε το χρόνο. Και με σχεδόν ευτυχία θα ήθελα να σας ξανα μεταβιβάσω την Προεδρία. Κύριε Κώστερ, θα μπορούσαμε εν συντομία να εξετάσουμε το σημείο 10. Μπορούμε όντως κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τίμερμανς στην πρώτη τελευταία συνάντησή μας δήλωσε ότι η Κομισιόν αποσύρει την νομοθετική πρόταση για την μεταρρύθμιση του δικαίου περί Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Διότι αυτή απαιτεί ομοφωνία. Και αυτή η ομοφωνία δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες. Εμένα μου φαίνεται πραγματικά μη ρεαλιστική η πιθανότητα να ξεκινήσουμε μια νέα πρωτοβουλία όσο και αν θεωρώ ότι έχει κάποια σκοπιμότητα το να φτιάξουμε ένα δίκαιο περί Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Κατέβαλα μια προσπάθεια με επιστολή προς τον κύριο Τίμερμανς να τον καλέσω να εγκαταλείψει την πρόθεσή του αυτή. Στην απάντησή του όμως ο κύριος Τίμερμανς μου δηλώνει ότι δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δίκαιο περί Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Επομένως, για την ώρα διαγράφεται αυτό το θέμα από το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται νομίζω να το σχολιάσουμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Άρα θεωρούμε ότι λύγει το θέμα αυτό. Αν όντω δεν έχετε αντίρρηση και δεν βλέπω κανένα να ζητεί το λόγο, τότε έχουμε δύο πολύ σύντομα πράγματα ακόμα και κλεισμένων των θυρών και όσοι παρακαλώ δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται ας αποχωρήσουν. Γρήγορα.